Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας γιατί έχουμε ήδη δύο σκιώδεις, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Οπότε, στην ημερήσια διάταξη έχουμε την εξέταση της, του σχεδίου γνωμοδότησης ε, Γιούνους Ομάρτζη για το Ταμείο Ενίσχυσης των Απόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λέγε, προφέρεται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματοποιήθηκε στην τελευταία μας συνάντηση Επιτροπής μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και γι' αυτό δεν θα επανέλθω, δεν θα επαναλάβω όσα τότε συζητήσαμε στο χώρο αυτό μια ανταλλαγή απόψεων με πολλά και διάφορα στοιχεία, αλλά παρακαλώ προσέξτε κάτι. Τι τι έγινε. Είχαμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις προτάσεις για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο και χαιρόμαστε γι' αυτό για ένα σχέδιο επιστημιστικής βοήθειας στους άπορους ε, και Όσον αφορά όμως τα διάφορα ποσά, ήταν 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι πολύ λιγότερα από όσα περιμέναμε, πολύ λιγότερα από τις ανάγκες πραγματικές, γιατί θα χρειαζόταν στις διάφορες οργανώσεις περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών. Και στη τελευταία μας συνάντηση το είπα, δεν θα το επαναλάβω, δεν θα επιμείνω, δεν μπορούμε πραγματικά να καταλάβουμε γιατί τώρα που έχουμε αυτή, αντιμετωπίζουμε αυτή την οξία κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απορεί όλο ένα και γίνεται μεγαλύτερος ο αριθμός τους γιατί αυτή η αντιμετώπιση και προσκληθήκαμε την ακρόαση του Βαντερποίτ του Προέδρου για το τι ακριβώς έγινε στο τελευταίο Συμβούλιο και μας είπε ο Πρόεδρος ότι δεν είχαμε μια μείωση σχετικά με το πρόγραμμα αυτό. Είναι όμως λάθος αυτά τα λόγια. Το γνωρίζετε ότι τα ποσά αυτά μειώθηκαν. Το 2010 είχαμε κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια. Μπορούμε να κάνουμε εύκολα τον υπολογισμό επί 7, αλλά λοιπόν είχαμε 3,5 δισεκατομμύρια. Και τώρα προβλέπονται 2,5 δισεκατομμύρια. Αλλά λοιπόν, αν το συγκρίνουμε με τον τελευταίο προγραμματισμό, έχουμε 1 δισεκατομμύριο μείων. Και ακόμα περισσότερο όμως ε, χρήματα λείπουν για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Ε, αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε ενώ ε, δεν ελέγχουμε την κατάσταση σε τον προπολογισμό. Και αυτό επί της αρχής ε, ποια ήταν η επιλογή μου. Να καταθέσω μία τροπολογία στην οποία λέω ότι θα πρέπει όσον αφορά τα ποσά αυτά να είναι στο ύψος των αναγκών για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες σε όλα τα κράτη-μέλη τα 27 κράτη-μέλη θα μπορούν να καλυφθούν από το ταμείο αυτό, κάτι που δεν συνέβαινε όμως τελευταίο προγραμματισμό. Εκεί συμπεριλαμβανόταν 20 ε, με 21 κράτη, τώρα και τα 27. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι αυτή. Να προχωρήσω στη δεύτερη. Χαίρομαι για την όλη κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έντονη κινητοποίηση από εμά με όλες τις πολιτικές ομάδες που συμμετείχαν για να διατηρηθούν αυτά τα ποσά και η κινητοποίηση και του Κοινοβουλίου και των πολιτών μπορώ να διαβεβαιώσω ότι έφεραν θετικά αποτελέσματα γιατί έτσι έχουμε να διαθέτουμε ένα νέο, μάλλον ε, θα πρέπει να συζητήσουμε ένα νέο κανονισμό Τίθεται τώρα θέμα στο νέο κανονισμό, ο οποίος προτείνεται όμως κάτω από δύσκολες συνθήκες και λόγω του χρονοδιαγράμματος της Επιτροπής Απασχόλησης ε, προσπαθούμε να υποβάλουμε προτάσεις ε, και είδαμε ποια είναι τα προβλήματα για να δούμε τι είναι επιλέξιμο Πότε ξεκίνησε αυτό το ταμείο, το χειμώνα του 85-86, πολύ σκληρός χειμώνας. Ξεκίνησε από την Επιτροπή Ροκάρ και ο στόχος ήταν να ανταποκριθεί στις ανάγκες τις επιτιστικές αυτά και μόνο και το συζητήσαμε στη τελευταία μας επιτροπή ε, εδώ αφορά όμως και την ε, διανομή κάποιου υλικού, διάφορου υλικού και όχι μόνο τροφίμων για τους άπορους. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να είναι με προϊόντα διατροφής ε, για να θρέψει κόσμο. Έτσι ξεκινάει η κοινωνική ένταξη κόσμου. Δεύτερη παρατήρηση μετά από τις συζητήσεις με τις ε, διάφορε ενώσεις που βοηθούν για την εφαρμογή των κανονισμών ώστε οι φιλανθρωπικές αυτές οργανώσεις ε, να μην επιβαρύνονται διοικητικά περισσότερο τώρα από ό,τι στο παρελθόν λόγω των νέων αυτών κονδυλιών. Δεύτερη σειρά τώρα προτάσεων, τις οποίες και διατυπώνω στην έκθεση αυτή και υπενθυμίζω ότι στα πλαίσια αυτής της βάσης που θα οργανωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μια σελίδα ίντερνετ κλπ και για τις ε, υπερφυριακές ε, περιοχές να μην λησμονηθούν αυτές και αυτή η ιστοσελίδα να απαριθμεί τις διάφορες ε, φιλανθρωπικές οργανώσεις που λαμβάνουν χρήματα. Έχουμε ένα προβληματικό σημείο. Είναι η κατάργηση της συγχρηματοδότησης. Δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά. Ήταν στο ύψος του 85% και προτείνω να είναι πια 100% γιατί δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα όλα τα κράτη-μέλη να καλύψουν το σύνολο, άρα λοιπόν ίσως αντιμετωπίσουμε καταστάσεις πραγματικά δύσκολες. Και επίσης διατυπώνω διάφορες προτάσεις, αλλά είναι περισσότερο συμπληρωματικέ. και θα ήθελα να ακούσω την άποψη των συναδέλφων για τα θέματα τα οποία συλλογίζομαι και τα οποία ξεκίνησαν και από συζητήσει με τις φιλανθρωπικές οργανώσεις αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι πρότεινα στην έκθεσή μου ότι η επιστημιστική βοήθεια που θα πρέπει να αποβλέπει σε υγιή τρόφιμα τη διανομή τους ε, ισορροπημένα και διάφορα. Η Ευρωπαϊκή όμως Επιτροπή με ενημερώνει ότι αυτό ίσως επιβαρύνει τις φιλανθρωπικές ε, οργανώσεις για να αποδείξουν ότι αυτά τα τρόφιμα είναι ισορροπημένα, διάφορα και υγιεινά. Αντιμετωπίζουν λοιπόν κάποιες δυσκολίες. Θα πρέπει να αποφασίσουμε και ελπίζω στα πλαίσια των ανταλλαγών απόψεων με τους συναδέλφους ότι θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε συγκεκριμένα για κάτι. Το δεύτερο που θα ήθελα να θέσω στους συναδέλφους είναι οι δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τη Eurostat. Ποιος θα λάβει υπόψη, τους, ε, υπόψη της Eurostat για να δει ποιος είναι πραγματικά ο, άπειρος, ο άπορος ε, πληθυσμός και ποιοι απειλούνται από τη φτώχεια. Θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι άποροι και από το 2009 και μετά δεν ξέρουμε αν αυτό επαρκεί. Χρειάζεται να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε μία απάντηση. Άλλο ένα θέμα για το οποίο χρειάζεται να τοποθετηθούμε είναι ο ορισμός της συχνότητας εργασίας συχνότητα εργασίας είτε επίπεδο αμοιβή. Είναι δύο διαφορετικοί ορισμοί. Με ανταλλαγές απόψεων με την Επιτροπή για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης, τι μας λέει η Επιτροπή. Αυτό το η συχνότητα μας επιτρέπει να δούμε καλύτερα τα πράγματα και να συμπεριλάβουμε και εκείνα τα νοικοκυριά που πραγματικά απειλούνται από τη φτώχεια αλλά και εδώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Βλέπετε ότι στην Επιτροπή περιμένω να ακούσω όχι μόνο ηχηρές δηλώσεις προθέσεων. Ε, πραγματοποίησα μια ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή πριν από κάποιο καιρό και είπαμε ότι αντιδράμε έντονα σε αυτό και χρειάζεται μια κάποια στιγμή βέβαια να συγγράψουμε μια έκθεση που να βοηθήσει στην βελτίωση του κανονισμού αυτού. Ελπίζω δε από τη συζήτηση αυτή και τις τροπολογίες που θα καταθέσετε θα έχουμε την ε, πληρέστερη πρόταση λεπτοδουλεμένη σε σχέση με αυτά που επιθυμούμε. Μια τελευταία παρατήρηση και τα είπαμε σήμερα το πρωί, ξεκινάει τώρα μια νέα διαπραγμάτευση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τον Προϋπολογισμό. Αυτό το θέμα της επιστημικής βοήθειας ε, τα τρόφιμα που θα διανέμονται θα είναι στο κέντρο των διαπραγματεύσεων. Το ελπίζω και ελπίζω επίσης ότι θα επιμείνει στη θέση του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα προπολογισμό που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών. Ε, αυτά προς το παρόν είναι τα πρώτα που θα ήθελα να επισημάνω και να σας πω ότι Είμαι έτοιμος να ακούσω κάθε υπόδειξη από τους συναδέλφους ώστε στο θέμα αυτό πάνω, όπως συμβαίνει άλλωστε από την αρχή, να διατηρήσουμε μια ομόφωνη, ισχυρή, δυνατή θέση της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Και τώρα η Μαρή Τερέζ Σμιθ από πλευράς Επιτροπής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ομαζή για το σχέδιο γνωμοδότησης. Συμφωνώ, έχουμε εισέλθει σε νέα περίοδο όπου χρειάζονται πραγματικές, ε, μάλλον ρεαλιστικές και συγκεκριμένες προτάσεις. Πρέπει να καθορίσουμε μια κοινή στάση που θα πρέπει στεναρά να υπερασπιστούμε και ενωμένοι. Όπως και εσείς, λυπάμαι που το Συμβούλιο στη συμφωνία του για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο υιοθέτησε πιστώσεις που θεωρούμε καθαρά ανεπαρκείς 2,5 η τελευταία πρόταση νομίζω ήταν 2,5 λοιπόν, ενώ οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ήθελαν 4 με 5 δις. Το σχέδιο προπολογισμού, όπως είπαμε, είναι, ε, ε, εξαρτάται τώρα τι, τι θα γίνει περαιτέρω θα ήθελα να χαιρετήσω την εργασία του εισηγητού και τις προτάσεις της τροπολογίας του. Προτείνει ε, και τέσσερα αλλαγέ ε, και οι συζητήσει τα ιδιαίτερα πλούσια στην τελευταία φορά. Καλό λοιπόν θα είναι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε ορισμένα σημεία πάνω αλλά οι τροπολογίες αυτές βέβαια είναι γεμάτες από καλές προθέσεις. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε και ποιες είναι οι πιέσεις του προπολογισμού. Φασίσαμε να δώσουμε μάχη για τον προπολογισμό, αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές. 5 δισεκατομμύρια στον προπολογισμό και χρηματοδότηση μάλλον και χρηματοδότηση 100% δραστηριοτήτων είναι κάτι ιδιαίτερα φιλόδοξο αλλά θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να υπερασπιστούμε παρόμοιε θέσει, γι' αυτό θα πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές, πραγματιστές ακριβώς, για να μην απογοητεύσουμε και τις φιλανθρωπικέ οργανώσει που έχουν δραστηριοποιηθεί και τις οποίες ε, υποστηρίζουμε και θα θέλαμε μια ενότητα. Ε, θέλουμε να δυνατό προπολογισμό, αλλά ταυτόχρονα με μια συγχρηματοδότηση εθνική, τα κράτη-μέλη χρειάζεται να λάβουν τι ευθύνε του όσον αφορά τι κοινωνικέ παροχέ και η νέα νομική βάση που και προτείνεται, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μα υποχρεώνει σε μια κοινή διαχείριση και επικορικότητα, την επικορικότητα ανάμεσα στα κράτη-μέλη κλπ. Εδώ η χρηματοδότηση είναι, έχει μια επιρροή, επηρεάζει τα πράγματα σαν μοχλός και θα πρέπει να δούμε και τις δυσκολίες στον προπολισμό των κρατών μέλων. Ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα συμβιβασμό το top-up να υιοθετήσουμε με 10 σημεία, 10 πόντους ακριβώς, να διατηρήσουμε τη χρηματοδότηση όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες τα κράτη-μέλη, τη χρηματοδότηση από εμά. Και επίσης ε, να δούμε τις δραστήριες οργανώσεις πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επενδυθούν των ε, ευθυνών τους και των ρεμοδιοτήτων στα πλαίσια αυτής της εταιρική σχέσης. Ε, έχουν κινητοποιηθεί για τον προπολογισμό και θα πρέπει να, παίξουν πάντα, να παίζουν πάντα ένα κύριο σημαντικό ρόλο. Αλλά κάπως λιγότερο να υποστηρίξω για τη φύση των ε, οργανώσεων που εταίρων μας ε, και ίσως ε, θα πρέπει να αφήσουμε τους οργανωτές να δουν πώς θα προχωρήσουν με το θέμα της επικουρκότητας με τα κράτη-μέλη. Και ακόμα να διευρυνθεί το πλαίσιο για τα είδη πρώτης ανάγκης πέρα από την επιστήμη βοήθεια καλή αυτή καθ' αυτή σαν ιδέα αλλά θα πρέπει ιδιαίτερα να επιμένουμε ότι για, τις για την προτεραιότητα αυτή, για την επιστημική βοήθεια, να καλύψουμε τι ανάγκες διατροφής αυτού του πληθυσμού που αντιμετωπίζει δυσκολίε. Ε, συμφωνώ με την τροπολογία για την απλοποίηση της όλης διαδικασίας. Ε, οι οργανώσεις οι οποίες έχουν δραστηριοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα είναι με θελοντική βάση. Δεν θα πρέπει να τους επιβαρύνουμε με γραφειοκρατικά, διοικητικά κλπ. Γιατί πολλές φορές οι κανονισμοί κοινοτικοί του υποχρεώνουν να αντιμετωπίσουν πολύ μα πολλή δουλειά. Και επίσης να διευρύνουμε την ε, βέλτιστη πρακτική με την κατάλληλη πλατφόρμα και επίσης το σελίδα για την πλατφόρμα αυτή και εγώ θα ε, καταθέσω τροπολογίες που θα υποστηρίζουν τη θέση του εισηγητού. Θα ρωτήσω μερικά πράγματα την Επιτροπή. Μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε και με γενικό τρόπο. Γιατί γίνεται, πόσα, πόσα θα πάνε ένα κράτος μέλος, τι γίνεται, με ποιο τρόπο καθορίζεται αυτή η κατανομή και θα παρθούν από το κοινωνικό ταμείο σε εθνικό επίπεδο. Πώς ακριβώς θα συνδυάσουμε μια ελάχιστη ε, επένδυση του κοινωνικού ταμείου με την κατανομή αυτή ανάλογα με τον πληθυσμό στον οποίο στοχεύουμε και επίσης ε, αυτά τα ποσά είναι και στα πλαίσια των κοινωνικών παροχών. Τι γίνεται, μήπως είναι όλα αυτά εις βάρος και της απασχόλησης. Πώς θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε τους σχετικούς στόχους ή αυτούς τους στόχους με το κοινωνικό ταμείο το οποίο είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ προσέξτε ότι θα μπορούσε να δοθεί ιδιαίτερα η πρόταση τη Επιτροπής. Ε, είναι νομικά ιδιαίτερα τομέα. τομέας. Γνωρίζουμε ότι διάφορα κράτη-μέλη δεν έχουν πιστεί ότι το ταμείο αυτό, το ποσό αυτό και οι δράσει του κοινωνικού ταμείου είναι κατάλληλε όσον αφορά την πιστική βοήθεια και είμαι πεπισμένη και ελπίζω και εσείς να συμμερίζετε την πεποίθησή μου. Θα πρέπει να εμφανιστούμε ενωμένοι και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για να μην δώσουμε τροφή σε όσους θέλουν να επανεκκουπήσουν την επιστική βοήθεια. Θα πρέπει όλοι μαζί, το παραλαμβάνω αυτό, θα πρέπει να εγγυηθούμε τη διατήρηση αυτής της βοήθειας στους άπορους, θα αποτελεί μεγάλη νίκη και θα πρέπει η κοινωνική δράση η δική μας να φαίνεται καθαρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, να βοηθάμε τους πολίτες που υποφέρουν από αυτή την ατελειωτή κρίση. Η κυρία Νταντσίλα από πλευρά Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, όλοι συμφωνούμε ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη έχει αυξήσει τον αριθμό των ατόμων που χρήζουν βοηθείες και που απειλούνται από την έσχατη ένδια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Γι' αυτό είναι σκανδαλώδες να διαπιστώνουμε ότι περικόπτεται σε τέτοιο βαθμό ο προπολογισμό για αυτά τα τόσο μειονεκτικά, τα άτομα που αντιμετωπίζουν τόσα προβλήματα. Έχει μειωθεί κατά πολύ ο προπολογισμό λοιπόν αυτό και το πρόβλημα είναι ότι οι πιο ενδεείς λοιπόν δεν έχουν καμία δυνατότητα πρόσβαση σε παρικέ και ποσοτικά και ποιοτικά φαγητό, διατροφή. Πάνω από 40 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν είναι σε θέση να φάνε κάθε μέρα πρωτεΐνες, είτε ζωικές είτε τις ε, ισοδύναμες φυτικές, ε, που να αντιστοιχούν στο επίπεδο που συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και 25 εκατομμύρια παιδιών επίσης κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 5,7 εκατομμύρια δεν έχουν καθόλου καινούρια ρούχα παίρνουν μόνο μεταχειρισμένα ρούχα από φίλους και συγγενείς και 4,7 εκατομμύρια δεν έχουν ε, τα κατάλληλα υποδήματα για το χειμώνα ή για το καλοκαίρι. Τα παιδιά αυτά που πάσχουν από τέτοιες ελλείψεις έχουν πολύ μικρή πιθανότητα ε, να τα πάνε καλά στην εκπαίδευση ή ε, να έχουν καλή υγεία και μεταγενέστερα διακινδυνεύει, δια, κινδυνεύει η να εχουν καλη υγεια και μεταγενεστερα διακινδυνευει δια η ένταξή του στην κοινωνία. Είναι η μελλοντική άνεργοι της Ευρώπης, για τους οποίους ανέργους ανησυχούμε τόσο πολύ ως Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να ανησυχούμε όλοι, και ως πολίτες και σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πρέπει λοιπόν να εξακριβώσουμε συγκεκριμένα ποιοι θα πρέπει να λάβουν αυτή τη βοήθεια, να κάνουμε τις αναγκαίες ε, έρευνες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως ε, τις δαπάνες αυτές. Όπως ξέρετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο 31.000 φορείς ασχολούνται με το πρόγραμμα αυτό, με 8.000 εργαζομένους και δεκάδες χιλιάδες ε, εθελοντές. Πολλοί από τους εθελοντές ε, λαμβάνουν και ίδιοι επιστηστική βοήθεια. Καταλαβαίνουν λοιπόν ποιες ανάγκες εξυπηρετεί αυτό το πρόγραμμα. Όλες οι οργανώσεις αυτές που πολλές από αυτές είναι οργανώσεις εθελοντών, μη κερδοσκοπικές, χρειάζονται απλοποιημένους κανόνες για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και χρειάζονται και απλό τρόπο διαχείρισης του προγράμματος. Ωστόσο, θα πρέπει να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει σε λειτουργία και ένα κατεπήγον ταμείο εάν η κατάσταση επιδεινωθεί ακόμη περαιτέρω ή εάν προκύψει μια κρίση που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Υποστηρίζω επίσης την ιδέα να χορηγήσουμε και τους αναγκαίους χώρους ε, για τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που δίδουν δωρεάν ε, τρόφιμα που είναι κοντά στην ε, ημερομηνία λήξης τους Ούτως ώστε αυτά τα τρόφιμα να πηγαίνουν στις τράπεζες τροφίμων για τους φτωχότερους πολίτες της Ένωσης. Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο αναφέρθηκε ο εισηγητής και ο σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ, θα πρέπει να είναι μια ανταπόκριση σε καταστάσεις κρίσης, να μας χορηγεί δηλαδή προϊόντα ποιότητας ε, για να διανύμουμε στους απόρους. Και παράλληλα, το πρόγραμμα διανομής τροφίμων για τους ε, πλέον απόρους είναι ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει την αποφυγή του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των πολιτών μας, μαζί με προγράμματα που διευκολύνουν την πρόσβαση ε, των πολιτών μας στην αγορά εργασίας. Διότι ε, όταν ε, οι ενδεείς αυτοί οι πολίτες βγουν από το σπίτι τους για να ψάξουν να βρουν ε, δωρεάν διανομή τροφίμων, έχουν μια δυνατότητα να βρουν και άλλους συμπολίτε τους να συζητήσουν και επειδή ακριβώς το 2013 είναι και το έτος των πολιτών, καταδεικνύουμε με αυτόν τον τρόπο ότι οι πλέον άποροι πολίτες της Ένωσης που χρειάζονται τέτοια προγράμματα βρίσκουν όντως ανταπόκριση. Τους δίνουμε έτσι μια δυνατότητα και να λάβουν βοήθεια και να αντιληφθούν την αλληλεγγύη της Ένωσης έναντί τους. Πρέπει λοιπόν σε αυτούς που ε, είναι αντίπαλοι του προγράμματος αυτού να ε, καταδείξουμε σαφώς ότι υπάρχουν πολλά άτομα που ακόμη έχουν ανάγκη την καθημερινή αυτή βοήθεια σε τρόφιμα. Θα υποβάλω τροπολογίες, έχω πολύ καλή συνεργασία. Με τον εισηγητή, η κυρία Χούσμονα δεν είναι εδώ. Θα ζητήσουμε την, ε, από την Καρίμ Ντέλη να μιλήσει τότε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρζέ για τον συνάδελφο, γιατί δείχνει καθαρά κάτι εδώ στην Επιτροπή. Την Ευρώπη που προστατεύει τους ε, πλέον άπορους σε ένα πλαίσιο όπου δυστυχώς υπάρχουν ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων που δεν καταλαβαίνουν την ε, κατάσταση αυτή δέ αποφάσεις πάνω σε μεγάλη σημασία θέματα για την Ευρώπη και εδώ υπάρχουν ε, επιπτώσεις και αυτά τα σύνορα, η γραμμή του απαράδεκτου έχει ξεπεραστεί, την έχουν υπερβεί εδώ στην Ευρώπη. Και θα ήθελα πάνω σε αυτό κείμενο να θυμίσω ότι είμαστε στα με τον προπολογισμό της επόμενης περίοδου προγραμματισμού, όπως προτείνεται από πλευρά Συμβουλίου. Δεν ξέρουμε στο και αν κάτι έγινε την τελευταία στιγμή, μια βελτίωση για τους πλεονάπορους. Το πως όμως αυτό είναι ανεπαρκές, αν το συγκρίνουμε δε με το σημερινό πρόγραμμα και αν καταλάβουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες του νέου ποσού αυτού που μας προτείνει με 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν τα καταφέρουμε και δεν μπορούμε να την κατάλληλη μάχη κατά των άπορων και των άστεγων εδώ μέσα αυτής τη επιτροπής, με τις πρότασεις επιτροπή μα στέλνει ένα μήνυμα καθαρό ότι έφτασε η ώρα να ε, δράσει κανείς και αυτό είναι και το καθήκον μας. Θα πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Και μας ζητάει να καταθέσουμε πραγματικές προτάσεις ο εισηγητής. Θα ήθελα να υποβάλω δύο προτάσεις ιδιαίτερης σημασίας. Εδώ στο κείμενο, μια διάσταση που μας αρέσει ιδιαίτερα σε μας οικολόγους. Αυτές τα... δηλαδή μια λυσίδα πώληση που να είναι βραχία με έτσι θα δώσουμε τη μάχη μας ε, καλύτερα, αποτελεσματικότερα και τους ντόπιους παραγωγούς θα ενισχύσουμε και επίσης τις εποχιακές καλλιέργειες, τη γη μας, ε, τις παραγωγές μας και θα δώσουμε τη μάχη μας κατά της ε, κλιματικής αλλαγής με αυτόν τον τρόπο με τα εμπορεύματα. Και γιατί το είπα ότι οι πλέον άποροι έχουν δικαίωμα σε μια υγιή διατροφή ποιοτικά υψηλής αξίας. Και αυτή είναι η πρώτη πρόταση. Πρόσβαση σε μια εταιρική σχέση κυρίως. Θα αναβεβαιωθώ ότι όλοι οι εταίροι θα συνεργαστούν από το ξεκίνημα του επιχειρητικού προγράμματος και οι ντόπιοι αγρότες και οι διάφορες ενώσεις και τα μπακάλικα που συμμετέχουν Ποιος είναι υπέρ της ένταξης των άστεγων. Ε, και βέβαια μία πρόταση θα ήταν η απλοποίηση. Είμαι κατά της συγχρηματοδότησης. Διάφορα κράτη και διάφοροι τις κατοκυβερνήσεων δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να θέσουν αυτό σαν θέμα με προτεραιότητα και για την αξία αυτή του, του προγράμματος και αν ισχύει αυτή η συγχρηματοδότηση θα μπορούσαν να πάρουν άμεσα αυτά τα χρήματα οι διαφερόμενοι. Άρα λοιπόν απαιτείται μια απλοποίηση πρόσβασης στα χρήματα αυτά. Να ολοκληρώσω δε, να πω ότι οι αξίες οι ευρωπαϊκές ε, τις οποίες υπερασπίζουμε είναι απλές πραγματικά. Απλές, πολύ απλές. Θα πρέπει να ζει αξιοπρεπώς ο καθές πολίτης δεν είναι φιλανθρωπικό πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα βοήθειας ε, στους φτωχότερους και αποτελεί ένα σύμβολο για το τι μας λείπει σήμερα. Αυτό κάνουμε. Αυτό που μας λείπει είναι η αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ. Ο Τζιμπλασάκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για την παρουσίαση που μας έκανε και έχω ορισμένα σχόλια. Και επίσης μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, νομίζω προς, ε, ότι προς το συμφέρον της ε, απλοποίησης της εφαρμογής ίσως θα ήταν ε, σκόπιμο το Ευρωπαϊκό αυτό ταμείο για την στήριξη των πλέον απόρων να ενταχθεί στο ενιαίο πλαίσιο στρατηγικής. Έτσι, η χρήση αυτού του ταμείου και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα μπορούσαν να εντάσσονται στο ίδιο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Και ερώτηση προς την Κομισιόν. Έχει γίνει καμιά αποτίμηση των αναγκών των ε, διαφόρων κρατών μελών. Τι πόρους θα απορροφήσουν από ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και αν ένα κράτος ε, δεν απορροφήσει τους πόρους που του αντιστοιχούν, θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια του επιχειρησιακού του ίδιου προγράμματος για άλλες ανάγκες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Α, όχι, συγγνώμη, υπάρχει ε, μακρύς κατάλογος. Γιάνν Όλμπριχτ. Όχι. Όχι, ωραία. Νίλσεν. Ε, έχουμε πολλά άτομα ήδη στο κατάλογο, αλλά προσθέτουμε και άλλα. Ευχαριστώ. Θα επιχειρήσω να είμαι σύντομο. Όταν κάναμε αυτή τη συζήτηση την προηγούμενη φορά, είπα ότι δεν μου αρέσει αυτή η πρόταση ευθύ εξ αρχή. Άρα δεν συμφωνώ με τον εισηγητή ούτε με την ομάδα μου. Να εξηγήσω λοιπόν γιατί. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε είναι να μεταθέτουμε το βάρος της ευθύνης μεταξύ κρατών μελών και ένωσης. Ίσως επειδή για 15 χρόνια έχω διατελέσει δήμαρχος στη Σουηδία. Στη Σουηδία η τοπική αυτοδιοίκηση είναι υπεύθυνη για τους ε, απόρους, για τους αστέγους. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να παράσχει σε όλους ε, ένα χώρο για να μπορέσουν να κοιμηθούν. Έχει αυτή την νομική υποχρέωση. Εάν ε, κάνουμε αυτά που προτείνονται, θα προκύψουν τα εξή. Πρώτον, για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, το πιο σημαντικό είναι η πρόσβαση στην απασχόληση. Η ανεργία προκαλεί τη φτώχεια. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και χρησιμοποιώντας, χρησιμοποιώντας το κοινωνικό ταμείο που το χρησιμοποιούμε τώρα για να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Αν τώρα αρχίζουμε να αφαιρούμε από το κοινωνικό ταμείο πόρους στις επόμενες χρονιές θα του πάρουμε ακόμη περισσότερα του κοινωνικού ταμείου άρα τα χρήματα αυτά ή θα τα αξιοποιήσουμε για να βοηθήσουμε την εξέβρεση εργασίας ή ε, θα τα δώσουμε για τους απόρους. Άρα είναι επικίνδυνη αυτή η παρέκκληση. Επίσης, στη Σουηδία, όταν δημιουργήθηκε αυτός ο νέος μηχανισμός, όταν θα δημιουργηθεί, οι, οι δήμαρχοι στη Σουηδία θα πούνε «Α, υπάρχει ε, ενωσιακή χρηματοδότηση, άρα εγώ δεν χρειάζεται να κάνω τόσο πολλά». Και αυτό είναι πρόβλημα. Να το ξανασκεφτούμε λοιπόν. Μακροπρόθεσμα θα ωφελήσει την Ευρώπη αυτή η προσέγγιση ή όχι. Έχω τις αμφιβολίες μου με βάση την εμπειρία μου από τη Σουηδία και το συζητήσαμε και στο κόμμα μας. Και επίσης ε, συζητώντας ποιος ε, φέρει την ευθύνη για διάφορα θέματα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας διαβεβαιώ ότι με τέτοιες προτάσεις οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα αρχίσουν να κάνουν λιγότερα. Ευχαριστώ. Ποιος άλλος? Η Κωνσταντσα. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω μία παρατήρηση επί της αρχής να κάνω. Ξέρω ότι συχνά έχουμε εκθέσει στα αγγλικά και διαβουλευόμαστε επ' αυτών. Πιστεύω 99% των συναδέλφων επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι το πρόβλημα των Αγγλικών. Όλοι γνωρίζουν Αγγλικά. Αλλά έχω μεγαλύτερε δυσκολίε όταν έχουμε θέμα διαβουλεύσεων στα γαλλικά. Δεν γνωρίζω αρκετά γαλλικά. Δεν μπορώ ούτε να τα διαβάσω, ούτε να τα μιλήσω, ούτε να διαπραγματευτώ ώστε με βάση ένα κείμενο να μπορώ να προχωρήσω έτσι στα γαλλικά. Δεν γίνεται αυτό. Και θα ήθελα εδώ να το πω, είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να μιλήσω για κάτι το, το οποίο δεν μπορώ να το διαβάσω. Μπορώ να το διαβάσω, δεν μπορώ να τα κατανοήσω όλα τέλεια. Αυτό είναι παρατήρηση επί της αρχής και νομίζω ότι δεν επιτρέπει να δουλεύουμε καλά και σωστά αυτού του είδους η διαδικασία να έχουμε σε άλλες γλώσσες κείμενα διαθέσιμα. Τουλάχιστον να είχαμε μια μετάφραση εργασίας, έστω στα αγγλικά, να ξέρουμε για τι πράγμα κάνουμε λόγο. Οι τροπολογίες μέχρι την Πέμπτη πρέπει να είναι έτοιμες, αλλά δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω μέχρι τότε με αυτούς τους όρους εργασίας. Αυτό πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν θέλουμε αυτό το πρόγραμμα και τα λοιπά. Έχουμε ξεπεράσει αυτού του είδους τις συζητήσεις. Αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πώς δημιουργήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Στον τομέα της πολιτικής για τη γεωργία ξεκίνησε. Όταν είχαμε βουνά βουτύρου από θέματα γάλακτος, ε, υπερπλεονάζοντα δηλαδή ποσότητες που πλεόναζαν. Και τώρα για την αντιμετώπιση αυτής της υπερπαραγωγής ε, θα έχει νόημα να δίνεται αυτό, αυτή η υπερπαραγωγή σε εκείνους που δεν έχουν ε, αυτή την ευημερία και χρειάζονται τρόφιμα λόγω του ότι υφίστανται τα πάνδυνα. Τώρα δεν έχουμε αυτού του είδους την υπερπαραγωγή και γι' αυτό υπήρξε η απόφαση να εξαιρεθεί, να βγει αυτό από την πολιτική ιδιοργία. Συζήτηση, χρειαζόμαστε αυτό το πρόγραμμα ή όχι και αν το χρειαζόμαστε πώς θα χρηματοδοτηθεί. Αποφασίσαμε πραγματικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα χρηματοδοτείται και το υποστηρίζω και ως πρόταση, ως πρωτοβουλία. Για εκείνες τις χώρες που δεν έχουν δυνατότητες οι ίδιες να αντιδράσουν και να κάνουν κάτι. Ουσιαστικά είναι αρμοδιότητα βέβαια των κρατών μελών. Και γι' αυτό ξέρω από την άλλη πλευρά ότι υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις και στην ίδια την Ομοσπονδιακή Γερμανία και στη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα οι Γερμανοί συνάδελφοι ήταν πολύ επιφυλακτικοί διότι θεωρούμε ότι κάπως ε, στοχεύει στην κατεύθυνση του Γένς, ε, αυτό που είπε ο Γένς. Δεν είναι δηλαδή αρμοδιότητά μας. Ωραία, περασμένα ξεχασμένα αυτά, αλλά να ξεκινήσουμε τώρα λέγοντας ότι πρέπει να αυξήσουμε τα κονδύλια, περισσότερα χρήματα να δίνουμε και όχι μόνο για τρόφιμα αλλά και επί παντός άλλου του επιστητού, νομίζω ξεπερνά την ουσιαστική θεμελιώδη ιδέα που είχαμε αρχικά. Δηλαδή να δώσουμε μια ευκαιρία συμμετοχή στην αγορά εργασία στους ανθρώπους που χρειάζονται κάτι τέτοιο. Το είπε ο Γιάννης μόλις πριν. Εμείς το ίδιο το μέσο, το εργαλείο αυτό, δηλαδή την συμπερίληψη, την ένταξη των ανθρώπων στην κοινωνία και στις, εργα... διαδικασίες για να βρουν θέση εργασίας, δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε και να μοιράζουμε ελεημοσύνες, να τους δίνουμε, ας το πω έτσι, ένα χαρτζιλίκι στο χέρι και τίποτα άλλο. Δεν είναι αυτό το νόημα της πολιτικής μας. Γι' αυτό ναι, για τους πιο φτωχούς, με συγκεκριμένα κριτήρια κριτήρια σε σχέση με τις χώρες ε, που ε, μπορούν να το διαθέσουν έτσι γιατί λόγω συγχρηματοδότησης ε, διότι ξέρω τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει αν αρχίσει να χρησιμοποιείται από εκείνους που δεν πληρώνουν δεκάρα. Είμαστε λοιπόν για αυτού του είδους τις αρμοδιότητες να χρηματοδοτηθούν όλα όσα κανονικά βρίσκονται στην ευθύνη των κρατών μελών. Αυτό πρέπει να είναι το κίνητρο, να σκεφτούν τι μπορεί να γίνει στο επίπεδο των κρατών μελών για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Παρακαλώ τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές σε σχέση με τις τροπολογίες να διασφαλίσουν ε, αυτή την πτυχή. Δεν μπορώ εγώ να συμμετάσχω υποβάλλοντας τροπολογίες γιατί έχω αυτό το γλωσσικό πρόβλημα που είπα πιο πριν. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Ντέλη που ζήτησε το λόγο, να σε ενημερώσω γιατί δεν υπάρχει μετάφραση. Ε, υπήρχαν ε, έκτακτες καταστάσεις. Παρά το ότι το ζητήσαμε, η Επιτροπή Απασχόλησης ε, αρνήθηκε να αναβάλει για την επόμενη συνεδρίαση την ψηφοφορία. Οπότε η μόνη δυνατότητα να συμπεριληφθεί η γνωμοδότησή μας ήταν να το συζητήσουμε τώρα. Οπότε δεν υπήρχε επαρκής χρόνος ούτως ώστε οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να μας στείλουν τις μεταφράσεις. Η έκθεση βεβαίως... Ε, η έκθεση είναι στα αγγλικά, λέει η πρόεδρος. Θα μπορούσαμε, αν θέλετε, να μην εγκρίνουμε την γνωμοδότηση ή να την εγκρίνουμε παρά τις γλωσσικές δυσχέρειες, παρά το ότι δεν έχουμε τις μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες. Δεν τις έχουμε τώρα εδώ εγκαίρως. Η ε, κυρία πάλι. Ευχαριστώ κυρία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, να πω στον Σουηδό συναδελφό μου να προσέξει λιγάκι. Όταν μιλάμε για φτώχεια και όταν λέμε οι θέσει εργασίας θα λύσουν το πρόβλημα, να υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ευρώπη εκατομμύρια φτωχούς που λαμβάνουν επιστημιστική βοήθεια και που έχουν θέση εργασίας. Η εργασία δεν, μας, δεν τους προφυλάσσει από τη φτώχεια. Μας λέτε ότι θα τους δώσουμε δουλειά για να μην είναι φτωχοί. Δεν επαρκεί. Εάν δεν αξιοποιήσουμε αυτό που ψηφίσαμε στην πλατφόρμα καταπολέμησης της φτώχειας, δηλαδή το ελάχιστο εισόδημα για όλους και όλες, δεν επαρκεί η απασχόληση πρέπει να θέσουμε το θέμα του ελάχιστου εισοδήματο. Και κάτι άλλο. Κάποιο είπε προηγουμένω, είναι θέμα αρμοδιότητα των κρατών μελών. Μα πώς θέλετε να δημιουργήσουμε την Ευρώπη που προστατεύει. Εγώ θέλω την Ευρώπη που προστατεύει, που χορηγεί περισσότερα δικαιώματα στους πολίτες της. Εάν τους πούμε στους πολίτες, κοιτάξτε, τα κράτη-μέλη, το καθένα θα φροντίσει για τους ε, απόρους του. Πού είναι λοιπόν η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό από πλευράς ε, συμβολισμού πρέπει να προκύψει από το κοινοβούλιο μας. Εγώ σκέφτομαι την Ευρώπη όπως ε, τη σκέφτονταν και οι ιδρυτικοί πατέρες που έλεγαν ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαιώματα. Και ένα από τα δικαιώματα είναι το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή. Αν εμείς που είμαστε οι πρέσβεις της Ευρώπης δεν έχουμε πλέον πια αυτές τις αξίες. Δεν θέλουμε να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, τότε φοβάμαι πολύ για την Ευρώπη του αύριο. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, να ζητήσω από το Γιούνους να κάνετε τελικά του σχόλια. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί μας επιτρέπει να καταλάβουμε επί της ουσίας τις θέσεις των μεν και των δε. Επιτρέψτε μου να πω ότι μου φαίνεται κάπως περίεργο να ακούμε να λέγεται ότι δεν είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Χρειάζεται να επενθυμίσω ότι στη συνθήκη της Ρώμης αναγράφεται το καθήκον προσφοράς σε όλους υγιεινή, ισορροπημένη και θρεπτική διατροφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο την εξάλληψη της ένδυας μέχρι το 2020. Είναι καθαρά ευρωπαϊκό θέμα και είναι καθήκον μας να αγωνιστούμε και σε αυτό το μέτωπο. Από τότε που ανέλαβα αυτή την έκθεση, λαμβάνω πάρα πολλά email. Ξεχυλίζει το ηλεκτρονικό μου γραμματοκιβώτιο. Ξέρετε ότι πολλές συζητήσεις μας δεν συγκινούν ε, τους πολίτες. Αλλά για το θέμα αυτό υπάρχουν υψηλές προσδοκίες και ενδιαφέρον από την κοινή γνώμη. Γιατί, όπως είπε και η Καρίμα, είναι πολύ σημαντική η συμβολική διάσταση. Ιδιαίτερα σημαντική. Σε αυτή τη συγκυρία διαπιστώνουμε όλοι την αυξανόμενη μεταξύ των πολιτών έλλειψη ικανοποίησης και δυσαρέσκεια με τους θεσμούς, δεν θα πρέπει να μην αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να διορθώσουμε αυτή την αρνητική εξέλιξη. Τέθηκαν ορισμένε ερωτήσει. Ορισμένε αφορούσαν ε, την Επιτροπή. Για αυτές που με αφορούν. Απλούστευση των διαδικασιών. Βεβαίως, Βεβαίως, μια σειρά από τροπολογίες που υπέβαλα επιδιώκουν αυτό το στόχο. Διότι εφόσον ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο εντάσσεται στη διαδικασία της πολιτικής συνοχής υπάρχουν οι αναγκαίοι έλεγχοι στους οποίους πρέπει να συμμορφούνται οι οργανώσεις αυτές και που δημιουργούν προβλήματα. Επίσης ε, συμμετέχουν περισσότερο οι περιφερειακοί φορείς και αυτό βασικό είναι ουσιώδες όλες οι οργανώσεις, όλοι οι φορείς να μπορούν να συμμετέχουν πολύ ενεργά στον καθορισμό των στόχων και επ' αυτού έχουμε υποβάλει τροπολογίες. Να διευκρινίσω επίσης Ήταν βέβαια ερώτηση προς την Κομισιόν, αλλά να διευκρινίσω. Οι χρηματοδοτήσεις ε, που θα χορηγηθούν στα κράτη-μέλη θα βγουν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και εδώ θα ήθελα να ακούσω την ε, απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνώ επίσης με την πρόταση της Καριμά για την αξιοποίηση των ε, τοπικών υψηλής ποιότητας προϊόντων. Βεβαίως, να το κάνουμε αυτό, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι οι φιλανθρωπικές οργανώσεις θα πρέπει να υφίστανται συμπληρωματικούς περιορισμούς που θα περίπλεκαν ακόμη περισσότερο τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν. Θα δούμε σε τι βαθμό είναι δυνατόν να υιοθετήσουμε αυτή την άποψη. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε εντελώ τη φύση της Επιτροπής της Κομισιόν. Θέλουμε η πρόταση αυτή να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ανάγκες των τραπεζών τροφίμων διότι όπως μας έχει προταθεί ο κανονισμός περιέχει μερικές ασάφειες που μπορεί να περιπλέξουν την κατάσταση. Τελευταίο, το είπα και στην αρχή, το δημοσιονομικό θέμα είναι το βασικό. Προφανώς όσο καλός και αν είναι ένας κανονισμός δεν θα παίξει κανένα ρόλο αν δεν επαρκούν οι πιστώσεις. Καλό λοιπόν να κινητοποιηθούμε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για να ε, καθοριστεί αλλιώς ο προϋπολογισμός. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Να αποφασίσουμε την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, πολύ σύντομη, 21η Φεβρουαρίου, 6 το απόγευμα. Οπότε λύγει το θέμα αυτό. Υποθέτω ότι μπορούμε να περάσουμε τώρα στο επόμενο, το 12. Λάμπερτ Φανίστελ Ρόι και Κωνσταντσε Κρέλ να μας ενημερώσουν για τις διαπραγματεύσεις για το γενικό κανονισμό. Ο κύριος Ρόε. Την προηγούμενη φορά οι συνάδελφοι μου είπαν ότι είπα πολλά. Οπότε τώρα θα είμαι πολύ σύντομος. Να μιλήσει πρώτα η Κωνσταντσα. Πρόεδρος. Παρακαλώ, η Κωνσταντσα. Οκ, θα μιλήσω λίγο περισσότερο, αλλά λίγο περισσότερο. Ευχαριστώ, Λάμπερτ. Μετά την προηγούμενη ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής κάναμε τρεις τριμερείς διαλόγους και σε σύγκριση με άλλους τριμερείς διαλόγους και άλλες επιτροπές έχουμε πολύ καλό ρυθμό. Ο επόμενος τριμερείς διάλογος είναι αύριο το απόγευμα. στις ε, συζητήσεις αυτές. Συζητήσαμε το παράρτημα του κοινού στρατηγικού πλαισίου. Αυτό ήταν αρκετά δύσκολο γιατί για ορισμένα σημεία διαπραγματευόμασταν πρόταση-πρόταση ενώ για άλλα τμήματα δεν υπήρχαν τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, αλλά να είναι σαφές ότι εμείς ήμασταν οι πρώτοι που προτείναμε κάτι. Γιατί προηγουμένως σας είχαμε πει ότι αποδεχθήκαμε το κείμενο του Συμβουλίου, αλλά μετά διαπιστώσαμε ότι το κείμενο του Συμβουλίου ήταν copy-paste του δικού μας. Έχουμε λοιπόν το κοινό το παράρτημα του κοινού προγράμματος του κοινού πλαισίου στρατηγικής και συζητήσαμε και το άρθρο που αφορά τα άρθρα 10, 11 και 12. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. πιο δύσκολη συμφωνία, ε, το πιο δύσκολο θέμα είναι αν θα υπάρξει κατεξοδότηση πράξη ή όχι. Όπως ξέρετε η Επιτροπή πάντα ζητάει μία εξουσιοδότηση πράξη ή το Συμβούλιο το απέρριψε ενώ εμείς είπαμε ότι για μας το κύριο θέμα είναι ο ίδιος ο κανονισμός. Και συζητάμε περαιτέρω για το θέμα της κατεξοδότησης πράξης. Αλλά δεν υπάρχει συμφωνία για το εάν θα υπάρξει ή όχι τέτοιου τύπου πράξη. Αυτό λοιπόν μένει να αποφασιστεί. Η Κομισιόν είπε ότι θα μας υποβάλει αναλυτική πληροφόρηση τι θα περιέχει αυτή η κατεξοδότηση πράξη και ελπίζω να μπορέσουμε να το συζητήσουμε αύριο στον επόμενο τριμερή διάλογο για να καταλήξουμε. Χθες τελειώσαμε το θυματικό κομμάτι που αφορά το εδαφικό τμήμα την ε, ανάπτυξη των ε, διαφόρων εδαφών και τις στρατηγικές για την τοπική ανάπτυξη και επίσης για τις ε, ομάδες τοπικής δράσης. Το μόνο θέμα που παραμένει είναι και πάλι εάν θα υπάρξει κατεξοδότηση πράξη για το 29, άρθρο 29 παράγραφος 6. Και εδώ η Κομισιόν θα καταρτήσει μία πρόταση. Ένα κομμάτι αυτού του τμήματος είναι πώς θα αναπτύξουμε τις περιοχές. Είναι το πρώην άρθρο 99. Τα επόμενα βήματα θα είναι το θεματικό τμήμα για την ε, εξάντε αιρεσιμότητα και για το πλαίσιο απόδοσης. Η εξάντα αιρεσιμότητα είναι λίγο δύσκολη γιατί δεν έχουμε κάποιο κείμενο βάση του οποίου να διαπραγματευτούμε. Είναι περίπλοκο θέμα και ελπίζω μέχρι την επόμενη Τετάρτη, αύριο 8 δηλαδή, να έχουμε μια πρόταση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και ελπίζω να προχωρήσουμε ταχαίως. Έχουμε λοιπόν όπως είπα κατακτήσει ένα καλό ρυθμό. Ο γενικός κανονισμός είναι βέβαια περίπλοκος. Άρα δεν τα πάμε και άσχημα, αρκετά γρήγορα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να υποβάλουμε το αποτέλεσμα στην Ολομέλεια πριν τις καλοκαιρινές διακοπές Οπότε αφήνουμε και αρκετό χρόνο στα κράτη-μέλη, τις περιφέρειες κτλ. να εκπονήσουν τα επιχειρησιακά προγράμματα. Αλλά εγώ προσωπικά και νομίζω ότι συμφωνεί και ο Λάμπερτ, θεωρώ ότι ορισμένες φορές είναι δύσκολο να διαπραγματευτεί κανείς με το Συμβούλιο που δεν είναι διατεθειμένο να πει ναι, ναι, έχετε δίκιο ή α, θα επανεξετάσω. Και τα θέματα αυτά είναι περίπλοκα. Όπως τα θέματα της αιρεσιμότητας. Ορισμένα δεν τα έχουμε συζητήσει ακόμη. Ελπίζω να βρούμε τρόπο να μπορέσουμε να καταλήξουμε στη συμφωνία και ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να είμαστε σε θέση να αρχίσουμε να συζητάμε τα επιχειρησιακά προγράμματα ούτω ώστε και οι ε, εταίροι μας περιφέρειες να δουν προς τα που πάει η συζήτηση. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη ενημέρωση. Και η Λάμπερτ, αν ξέχασα κάτι, παρακαλώ. πρόεδρος, ναι, εάν του δώσω το λόγο, λέει ο πρόεδρος. Ε, Λάμπερ, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Αν θέλετε οπωσδήποτε μόνο, ε, τέτοιες προσκλήσεις ε, δεν πρέπει να τις αρνείται κανείς. Απόλυτα σωστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και σπουδαία προβλήματα να επιλύσουμε. Η μακρο, για τη μακροοικονομική διάσταση οι και για τις επιδόσεις και έχουμε και την απόφαση του Συμβουλίου της προηγούμενης εβδομάδας. Αν δείτε αυτού του είδους τα θέματα πρέπει να δούμε τα ποσά τα οποία θα απαιτηθούν. 7% τι θα είναι. Ίσως καμιά φορά έχουμε αυτή την ε, αναδραστική πληροφόρηση, την ενημέρωση. Καμιά φορά υπάρχει και η ανάγκη να προβάλλουμε κάτι προς το μέλλον ως ε, πιθανότητα. Αν πάντα λέγεται το όχι, όχι και πάλι όχι, ε, τότε πώς μπορεί αυτό μέσα σε μια περίοδο 7 ετών να λειτουργήσει, να προβλέψουμε την έκβασή του, αλλά θα πρέπει να μην έχει γραφειοκρατική διεργασία και επιβάρυνση, δηλαδή απλά να δοθούν χρήματα με ένα γραφειοκρατικό τρόπο και να νομίζουν ότι επιλύονται τα προβλήματα. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε μια τέτοια, ας το έτσι, προοπτική στην ε, χρονική αυτή διάρκεια και να δούμε τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της προσέγγισης του Κοινοβουλίου, της προσέγγισης αυτών των θεμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο. Και θα πρέπει και στη συζήτηση να μπορέσουμε, όπως και στο Στρασβούργο, να δούμε τι μπορεί να επιτευχθεί. Ο κύριος Σάντορ να έρθει να υποβάλει κάποιες ιδέες, να υποβληθούν ιδέες και να προχωρήσουμε. Διαφορετικά θα κολλήσουμε. Δηλαδή σε σχέση με την ευελιξία, τι θα γίνει. Είναι δύσκολο να υπάρξει μια συμφωνία αν όλα αυτά δεν ενταχθούν. Καμιά φορά λοιπόν αν μπορούμε να έχουμε κάποιες ιδέες, να δούμε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιστεί, να προσεγγίσει, να έρθει προς τη δική μας πλευρά. Ίσως θα μπορούσαμε έτσι να είχαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αν δεν κινητοποιηθούν, ποιος ξέρει στο τέλος το τι θα απογίνει. Και θα πρέπει με το ε, Συμβούλιο να δούμε τι θα πρέπει να γίνει και σε σχέση και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα είναι δυσαρεστημένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συνάδελφοί μας από την Κοινωνική Επιτροπή πώς θα πρέπει, πώς θα κινηθούμε, πώς θα σημειωθεί κίνηση. Ναι, είναι ένα ερώτημα το οποίο θέτω. Εσείς μου δώσατε τον λόγο, δεν ήθελα να δημιουργήσω πρόβλημα. Ευχαριστούμε Λάμπερτ πολύ από τους σκιώδεις τώρα, από την ομάδα των σκιωδών εισηγητών. Θα ήθελε κάποιος να παρέμβει. Ο εσείς, ο κύριος Αματζή παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ. Δύο ειδών παρατηρήσεις. Ε, σήμερα το πρωί στη συζήτηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών τι είπα. Ότι Κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή συνθέτουμε την ομοθεσία σε θέματα συναπόφασης. Γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουμε ώστε τα όσα ζητούνται από το Κοινοβούλιο να γίνουν σεβαστά. Θα επιστρέψω λοιπόν και θα πάω στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα ήθελα δε των ε, συνεισηγητών να έχω την άποψή τους για το περιθώριο που έχουμε ακόμα έλιγμων στην εν λόγω διαπραγμάτευση. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρεται καθαρά, σαφώς αυτή η πιθανότητα η μακροοικονομική και ε, με αποθεματικά κλπ. Εδώ, τι θέλω να πω εγώ, τι έχουμε ακόμα. Και από τη στιγμή που όλα έχουν ε, εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο και αν η αρχή της συναπόφασης γίνεται σεβαστή. Δεύτερη παρατήρηση και ερώτημα μάλιστα στον εισηγητή είναι η δική μας η εντολή για τις διαπραγματεύσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την εντολή και παρακαλώ διορθώστε με αν κάνω λάθος. Δεν προβλεπόταν κάποιο κεφάλαιο για τη συνοχή των πέντε ταμείων με τη στατική του 2020 και την οικονομική ευρωπαϊκή διαχείριση. Αλλά τι γίνεται από το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων στον τριμερή αυτό διάλογο. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο τι κάνουν. Βλέπουμε ότι εξετάζουν τη στατική του 2020 με τον τρόπο του εξαμήνου του Ευρωπαϊκού πώς ε, συμμετείχαμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και το Συμβούλιο και η Επιτροπή κάθε φορά επανέρχονται με αυτό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και να σας πω κάτι ποια είναι η θέση μου, ότι είμαι αντίθετος και από τον εισηγητή τι τους ζητητές τη ζητάω την άποψή τους και ταυτόχρονα τους ζητήσω να μην απομακρυνθούμε από τη θέση μας και την εντολή που έχει οριστεί. Και εδώ το ξεκίνημα και νομίζω ότι συμμερίζεται αυτή την άποψη για την ε, πολιτική συνοχή. Δεν θα πρέπει αυτό να νερώσει με αυτή την αυστηρή λυτή ε, ρίση που μπαίνει εδώ σε αυτό το διατακτικό. Σας ευχαριστώ. Uh, Θα ήθελα μια πολύ σύντομη ερώτηση να αναφέρω μια πρωτοβουλία κοινοτικού επίπεδου Είχαμε και μακρότερες συζητήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση, τη δομή και το κόστος. Αν συζητήθηκε όχι δεν μπορώ να το πω, αλλά ο ειδικό τρόπος διοργάνωσης κοινωτικών πρωτοβουλίων που κατά λάθο θεωρείται ότι σε σχέση με τη CEP, την ΚΑΠ θα μπορούσαν να παρατείνουν ή και να διευρύνουν το πλαίσιο ε, για τη, από πλευράς του Λίντερ για την ανάπτυξη των ε, αστικών κέντρων, των πόλεων είναι ο τρόπος ε, λειτουργίας για αυτές τις δράσεις από το leader και υπάρχει και μεγάλο κόστος ε, λειτουργικών δαπανών υψηλό ποσοστό που δημιουργεί πολλές αμφιβολίες μήπως είναι υπερβολικά υψηλό όσον αφορά τις δαπάνες αυτές για να επικεντρωθεί κανείς στις δράσεις για τις πόλεις, για τα αστικά κέντρα. Για την περιοχή της ε, Υπέθρου εντάξει αλλά για τα αστικά κέντρα δεν είμαι τόσο βέβαιος αν αυτό αξίζει ή όχι με τέτοιες δαπάνες. Και δεύτερο, να δούμε αν συμβαίνει αυτό ή όχι. Πρόκειται για το ITI που συμπεριλαμβάνει το πρόβλημα της αντιπροσωπείας η αντιπροσωπεία έχει στεναρή αντίσταση από πλευρά του Συμβουλίου αλλά από πλευρά του ITI να συνεπάγεται αυτό την χρήση αντιπροσωπείας ή υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική δυνατότητα. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θα ήθελε να λάβει τον λόγο προτού δώσω τον λόγο να παρέμβουν οι συγητές η Κωνσταντσε Ιω Λάμπερτ η Κωνσταντσε πρώτη να σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας θα έλεγα Κάθε φορά καθίστατο απόλυτα σαφές ότι μια απόφαση από πλευρά Συμβουλίου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το MFF, και με μέρος της διαδικασίας συναπόφασης για την πολιτική συνοχής είναι μια εντολή προς το Συμβούλιο αυτό και υπό την Κυπριακή Προεδρία και υπό την Ιρλανδική Προεδρία και την Δανέζικη προηγούμενα κάθε φορά καθίστατο σαφές ότι μάλιστα πρόκειται απλά και μόνο για μια εντολή. Δεν θα θίξουμε καθόλου την διαδικασία συναπόφασης Πολύ με ενδιαφέρει να δω πώς θα μπορέσουν να επιλύσουν αυτό το δίλημα, αυτό το πρόβλημα και πώς θα καταλήξουμε σε μια θετική καλή απόφαση. Το μέλλον θα το καταδείξει αυτό. Δεν είναι πιο εύκολα τα πράγματα τώρα. Από την άλλη πλευρά όμως έχουν η λιμένη θέση εκείνη, έχουμε εμείς δικές μας θέσεις, πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μεταξύ μας. Όμως η εντολή για την διαπραγματευτική ομάδα είναι απόλυτα σαφής, έτσι δεν είναι. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τότε θα πρέπει να επανέλθουμε, να επιστρέψουμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή εδώ, να το συζητήσουμε αν μπορέσουμε να το επιλύσουμε πολύ καλά. Διαφορετικά θα πάμε στην Ολομέλεια θα προστρέξουμε ώστε το σύνολο του Κοινοβουλίου να εξεύρει μια λύση. Αυτή είναι η κατάσταση. Κάπου πρέπει να ληφθεί μια απόφαση, να λαμβάνεται απόφαση. Και ελπίζουμε ότι τα προβλήματα θα μπορέσουν να επιληθούν προηγούμενα, πρωτού καταλήξουμε στην Ολομέλεια αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε τις διεργασίες και τις διαδικασίες από πλευράς Κοινοβουλίου για να εξυπηρετηθούμε και να βρούμε μια λύση. Για το άλλο θέμα, ναι, συζητήσαμε όλα αυτά τα ζητήματα σίγουρα στον τριμερή διάλογο, ιδιαίτερα εχθές. Και για την ανάπτυξη της Υπέθρου, για τους χώρους της Υπέθρου, πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχή της μεθοδολογικής προσέγγισης από πλευράς ε, του leader. Και όσον αφορά τις δυνατότητες να επικεντρωθούν σε αστικά κέντρα στις πόλεις, μπορεί να γίνει αυτό από τα κράτη-μέλη, διότι έχουμε θετική πείρα, θετική εμπειρία. Αν θέλουν αυτή την αρχή μεθοδολογικά να την υιοθετήσουν και να την χρησιμοποιήσουν για άλλου είδους τέτοια σχέδια, προγράμματα, μπορούν να το κάνουν. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα, δεν, είναι, δεν επιβάλλεται κάτι τέτοιο δεσμευτικά. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αφορά τις κατηγορίες περιφερειών. Πώς αυτή η αρχή θα μπορέσει να συγκλίνει σε σχέση με τις πόλεις. Υπάρχει ένας ορισμός, προσδιορισμός που προτείνεται από το Συμβούλιο μια τέτοια περιοχή να έχει 10.000 μέχρι 150.000 ε, όσον αφορά τους κατοίκους. Υπάρχουν όμως πόλεις που είναι πολύ μεγαλύτερες, έτσι δεν είναι και υπάρχει και η δυσκολία ε, κατηγοριοποίησης. Υπάρχει το πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν προτείνεται μια διεργασία όσον αφορά το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την επίλυση του προβλήματος. Μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την ιδέα, αλλά να μην είμαστε δίσκαμπτοι, να μην δημιουργηθεί δισκαμψία στη λειτουργία, στη λειτουργικότητα αυτών των ε, προτάσεων. Και έχουμε και την ιδέα τώρα από την άλλη πλευρά που παρουσιάζεται να βελτιωθεί η δυνατότητα επιδόσεων και η, να χρηματοδοτηθεί η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας να μπορούν να εργάζονται και να χρησιμοποιήσουν τέτοιες στρατηγικές οι κάτοικοι αυτών των περιοχών Αναμένουμε ακόμα ένα άλλο συμβαστικό κείμενο ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να επιλύσει αυτά τα ε, προβλήματα. Υπάρχει αυτή η ιδέα όσον αφορά αυτή την προσέγγιση αλλά όχι η τελική διατύπωση του κειμένου. Πρέπει να δούμε λοιπόν και ποιο θα είναι και το κόστος ε, για να μπορέσει να επιτευχθεί μια τέτοια λύση. Από πλευρά των ITIs γνωρίζετε ότι είναι μια απόφαση των κρατών μελών να χρησιμοποιηθεί αυτό το μέσο ή όχι. Από τα κράτη-μέλη εξαρτάται και για τις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο του ITI μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν είναι υποχρεωτικά όλα αυτά, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θέμα μεθοδολογικό για την ανάπτυξη των τοπικών αυτών περιφερειών. Δεν είναι υποχρέωση, είναι ανοιχτό για να εφαρμόζεται η ελαστικότητα για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο Λάμπερτ. Μία ερώτηση που κάπως ε, μας κάνει να προβληματιστούμε ευρύτερα για αυτά τα οποία συνέβησαν τις προηγούμενες εβδομάδες και πώς θα πρέπει να δράσουμε ως Επιτροπή των Περιφερειών γενικότερα προσεγγίζοντας το όπως ε, παρακολουθώντας τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την ε, Σύνοδο Κορυφής στο τέλος τέλος η πολιτική συνοχής πήρε κάποια δισεκατομμύρια παραπάνω για να μπορέσει να προχωρήσει αλλά σε σχέση με τις περικοπές βλέπουμε ότι γίνονται περικοπές ε, στους τομείς μας και κανείς δεν είναι στο τέλος ε, ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Ας συνεχίσουμε να δούμε τι θα γίνει και το δεύτερο είναι το τι έγινε για παράδειγμα σε σχέση με την έρευνα και την ανάπτυξη υπάρχουν ε, φωνές που εκφράζουν αντιρρήσεις αν δείτε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις ήμουνα σε μια αντιπροσωπεία την προηγούμενη εβδομάδα και μπόρεσα πραγματικά να παρακολουθήσω τους ε, όσους παρενέβησαν και είπαν εντάξει, δεν είναι τόσο αρνητικά τα πράγματα όσο προσδοκούσαμε. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο τι στοχεύει να πει, τι σημαίνει, αλλά για την Ήτρε και τι προσπάθειες που έγιναν εντός και εκτός προϋπολογισμού είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτές τις συζητήσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπαν. Τι είπαν. Είπα τώρα διαπραγματευόμαστε και τώρα χρειαζόμαστε λοιπόν και τη δική σας συνεισφορά για αυτά τα οποία δόθηκαν για να υπάρξει μια ε, υπαναχωρώντας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην κοινωνία της γνώσης και της ε, αποτελεσματικότητας τώρα πρέπει να τηρηθούν όλα αυτά τα υπεσχημένα και να λειτουργήσουν σωστά και γίνονται διαπραγματεύσεις στους τριμερείς διαλόγους. Και τίθεται το ερώτημα, είναι η θεματολογική επικέντρωση, η επικέντρωση στη γνώση, η ευφυής εξειδίκευση, όλα αυτά κατοχυρώνονται μέσω των κανονισμών και των διατυπώσεών τους. Ελπίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό, αλλά δεν είμαι και τόσο βέβαιος, διότι κάποια πρέπει να ενταθούν σε έναν, στον κανονισμό με έναν τελικό τρόπο, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά και να συντονιστούν. Και εκείνοι οι οποίοι ε, ως γραφειοκράτες ε, θα πρέπει να ε, καθορίσουν τη ροή των κεφαλαίων δεν θα πρέπει να τροχοπεδίσουν τις εξελίξεις προσβλέποντας τις επόμενες διαπραγματεύσεις σε σχέση με το Κοινοβούλιο για παράδειγμα για το ότι θα πρέπει λόγω των κονδυλίων, λόγω των ιδίων πόρων και λόγω όλων αυτών των στοιχείων δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι και για την έλλειψη της καινοτομίας. Κατά κάποιο τρόπο πρέπει να δείξουμε και να αντισταθούμε σε όλα αυτά ότι εκ των κάτω προς τα άνω από την επικουρικότητα, από τις, ε, την εταιρική σχέση ε, για την ανάπτυξη θα πρέπει να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά και να δώσουμε τα κίνητρα για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Βλέπουμε ότι οι κλιματικές αλλαγές σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν τεράστιες επιπτώσεις. Το να συμπεριληφθούν τώρα αυτές οι πτυχές ε, όσον αφορά και την επικέντρωση για τα θέματα παιδείας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να υιοθετήσει μια ομένη άποψη για το τι πρέπει να γίνει σε σχέση με τα αποτελέσματα. Όχι να λέμε για το ένα α να υπάρχουν αντιρρήσεις, για το ένα β να μην είναι όλοι βέβαια απόλυτα ικανοποιημένοι, αλλά να δούμε ποιες ε, πτυχές υπάρχουν που από πλευράς του προϋπολογισμού μπορούν να διασφαλιστούν Υπάρχουν εδώ τα θέματα των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό. Εμείς έχουμε τα χρήματα αυτά τα οποία ε, πρέπει να δείξουμε στους άλλους εμπλεκόμενους ε, ότι η πολιτική την οποία ζητούμε να ακολουθήσουμε ως Κοινοβούλιο θα είναι ε, εκείνη η οποία απαιτείται και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για το Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής να εξυγχρονιστούν τα πράγματα, να αλλάξουν τα πράγματα και να βελτιωθούν γιατί διαφορετικά θα επαναλαμβάνει το Κοινοβούλιο τις θέσεις του ΕΣΑΗ. Λοιπόν, δύο μηνύματα. Το πρώτο θα μπορούσε να είναι ότι θα έπρεπε να δώσουμε προσοχή και να συνέρθουμε ως εισηγητές ε, με τα πέντε ταμεία υπό το πλαίσιο αυτού του κανονισμού να δούμε πώς θα μπορέσει να σημειωθεί πρόοδος και όλα αυτά να ενταχθούν σε μια σωστή αναλογία ε, στοιχείων και να συνέρθουμε επίσης και με τους εισηγητές για το Horizon για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Καινοτομίας ε, και Τεχνολογίας βλέποντας το τι γίνεται εκεί για παράδειγμα σε σχέση με την περιφερειακή ανάπτυξη ή την ε, ε, κοινωνία της ε, προηγμένης γνώσης. Ακριβώς τα ίδια συμβαίνουν εκεί όπως και με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θεματολογική επικέντρωση σε κάποια θέματα. Θεματολογική επικέντρωση ώστε να μπορέσουμε από την Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο να εστιαστούμε και να λειτουργήσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Να δούμε λοιπόν και για τον δικό μας κανονισμό και για τον κανονισμό έρευνας και ανάπτυξης να συντονίσουμε τα πράγματα να είμαστε πιο αποτελεσματικοί να τα κάνουμε όλα αυτά επικοινωνώντας σωστά ο ένας με τον άλλον. Γιατί διαφορετικά είναι πολύ δύσκολο να καταλήξει κανείς σε μια συζήτηση που επαναλαμβάνεται κυκλικά, τα επιχειρήματα ακολουθούν το ένα το άλλο αλληλοδιάδοχα σαν ένα δίσκο γραμμοφώνου. Μπορεί αυτό να αναπτυχθεί διαφορετικά. Αν στο τέλος το κοινοβούλιο για παράδειγμα, εγώ υποστηρίζω την ιδέα να δεχθούμε έστω και με πολλές αλλαγές ένα τέτοιο προϋπολογισμό για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αλλά πρέπει να δείξουμε, να καταδειχθεί ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα για το Περιφερειακό Ταμείο, το Ταμείο ε, περιφερικής Ανάπτυξης, ε, κοινωνικό ταμείο και το, ε, τους προϋπολογισμούς ε, για τις δράσεις αυτές. Δεν ξέρω πώς θα γίνουν όλα αυτά, αλλά αυτά πρέπει να εξετάσουμε σε ένα τέτοιο συντονισμό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό για σας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε σας. Και πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε τώρα στη δεύτερη έκθεση που θα είναι του Γιάν Ολμπριχτ. Παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ. Και εμείς προσπαθούμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Είχαμε τριμερή διάλογο 31 Ιανουαρίου και στις 18 Φεβρουαρίου κάναμε μια τεχνική συνάντηση. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που ήδη έχουν εγκριθεί από τα τρία θεσμικά όργανα, ενώ άλλα παραμένουν εκκρεμή. Πρώτον, υπάρχει προσωρινή συμφωνία για την επέκταση του εύρους ενίσχυσης Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις, θα θυμάστε. Υπάρχει προσωρινή συμφωνία ότι για την έρευνα, την καινοτομία, την, την ε, ε, ενεργειακή ε, αποδοτικότητα και την τεχνολογία πληροφόρησης και επικοινωνιών θα υπάρχει ευρύτερη χρηματοδότηση. Επίσης, προσωρινά συμφωνήθηκε να υπάρχει δυνατότητα να δίνονται χρηματοδοτήσεις για τις υποδομές στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και την επιλεξιμότητα μικρής κλίμακας προγραμμάτων στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού. Ε, συζητάμε ακόμη τι είπα να πει μικρής κλίμακας. Δεν ξέρω τι σημαίνει μικρής κλίμακας για το Παρίσι. Ξέρω τι σημαίνει μικρής κλίμακας για μια μικρή χώρα. Μικρής κλίμακας λοιπόν πολιτιστικές και τουριστικές υποδομές. Παραμένει ανοιχτό το θέμα της επιλεξιμότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων αναψυχής. Εδώ η Κομισιόν και το Συμβούλιο είναι ιδιαίτερος κατά. Καταφέραμε να καταργήσουμε την ε, ε, εξαίρεση των ε, υποδομών, στον τομέα των μεταφορών, τη πληροφορική κτλ. για τις πιο αναπτυγμένες περιοχές. Αυτό συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο, σημαντικό είναι αυτό. Συμφωνούμε λοιπόν για ορισμένα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι οι υποδομές για τις βασικές υπηρεσίες, αλλά αφού το καταργήσαμε δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Ο επόμενος τριμερής διάλογος θα αφορά αυτό το άρθρο. Πολύ σύντομα λοιπόν ελπίζω να κλείσουμε τη συζήτηση για το άρθρο 3 όσον αφορά τις προτεραιότητες για τις επενδύσεις. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που συμφωνήσαμε να προσθεθούν. Για παράδειγμα, ηλεκτρονικός πολιτισμός ή πολιτισμός, επιλεξιμότητα προγραμμάτων που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση για τα διάφορα είδη επιχειρήσεων, όχι μόνο μικρομεσαίες, αλλά κάθε επιχειρήση. Αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα και επίσης η κινητικότητα στις αστικές περιοχές. Έχει προσθεθεί στη θεματική συγκέντρωση μετά από πρόταση του Κοινοβουλίου. Να σας υπενθυμίσω ότι το επίπεδο της ενεργειακής απόδοσης ανεβαίνει στο 12% αναφορά και το Ταμείο Συνοχής. Η επιλεξιμότητα επίσης προγραμμάτων για την συμπαραγωγή ενέργειας και θέρμανσης. εφόσον είναι υψηλής αποδοτικότητας για τις ε, επενδυτικές προτεραιότητες θα συζητήσουμε την επόμενη φορά, αυτή τη βδομάδα δηλαδή. Τρίτον, η αστική διάσταση. Εντάσσεται στο γενικό κανονισμό, γιατί αφορά εταιρικές συμφωνίες με ποια κριτήρια, με ποιους ε, κανόνες θα επιλέγονται οι αστικές περιοχές. Εμείς ε, προτιμάμε λειτουργικούς ορισμούς, ενώ εκείνοι προτιμούν γενικά αστικές περιοχές. Υπάρχει θέμα ουσίας, δεν είναι μόνο θέμα διατύπωσης. Πιστεύω όμως ότι θα συμφωνήσουμε πάνω κάτω. Τι σημαίνει ανοιχτό. Αυτή είναι η ερώτησή μου και στην Κωνσταντσε τι, σημαίνει, τι είναι ακόμη ανοιχτό. Μιλάμε για αυτό το περίφημο 5%. 5% του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που αφορά τις ολοκληρωμένες αστικές δράσεις. Το πιο σημαντικό σε αυτό το 5% ποια είναι η προστιθέμενη αξία για την Κομισιόν που κάνει αυτές τις προτάσεις. Για αυτούς το πιο σημαντικό είναι, είναι η παραχώρηση ορισμένων στοιχείων ορισμένων αρμοδιοτήτων στις αστικές αρχές, όχι μόνο τις τοπικές, αλλά γενικά τις αστικές αρχές. Εμείς θελήσαμε να υπάρχουν διαφορετικοί ρυθμοί, διαφορετικά επίπεδα χορήγης αρμοδιοτήτων, εκχώρης αρμοδιοτήτων. Θα μπορούσε δηλαδή να έχουμε απλώς αρμοδιότητα που να εκχωρείται για την επιλογή προγραμμάτων μέχρι την πλήρη εκχώρηση που αφορά τη χρηματοδότηση συνολικά. Το Συμβούλιο δεν θέλει να εχωρίσει καθόλου αρμοδιότητες. Αυτό το θέμα παραμένει ανοιχτό. Η εντολή από την Επιτροπή μας είναι να προωθήσουμε την εκχώρηση αρμοδιοτήτων, ούτω ώστε να είναι πιο υπεύθυνε οι αστικές αρχές για τη διαχείριση των προγραμμάτων έναντι της διαχειριστικής αρχής. Αυτά είναι τα ανοιχτά θέματα Ευχάριστα με εξέπληξε το ότι η Επιτροπή Περιφερειών με ευχαρίστησε που υποστήριξα την ε, πλατφόρμα αστικής ανάπτυξης, αστικής αναγέννησης. Η Επιτροπή μας ήταν κατά, υπενθυμίζω. Αλλά η Επιτροπή μας εξήγησε ότι αυτό που προτείνει δεν είναι μια νέα πλατφόρμα όπως η πλατφόρμα 2020, αλλά προτείνει μια τεχνική πλατφόρμα για να ελέγχουμε εάν λειτουργούν ή όχι τα πιλωτικά προγράμματα. Είναι τεχνική ανταλλαγή πληροφοριών δηλαδή για το πώς προχωράει το κάθε έργο. Αλλά παρόλα αυτά η Επιτροπή μας έχει αρνητική εντολή δόση, άρα πρέπει να αλλάξουμε αυτή την αρνητική εντολή επανερχόμενη στην Επιτροπή, ενώ η Επιτροπή Περιφερειών θα το δεχόταν αν συνδεθεί με την Επιτροπή Περιφερειών. Δηλαδή, αν η Επιτροπή Περιφερειών συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, θα το αποδεχθεί. Αντίθετα, οι διάφοροι φορείς, οι Ευρωπόλεις και τα λοιπά και το πρόγραμμα Airbact είχαν πολύ ακραία άποψη στην αρχή αλλά το airbag είναι ε, σχετικά αυτόνομο αυτή τη στιγμή. Αν μπει σε αυτή την πλατφόρμα θα γίνει υποχείριο της Κομισιόν, υπηρεσία της Κομισιόν. Άρα πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει κατανοητό περί τίνος πρόκειται. Είναι πολύ ισχυρή η θέση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρκετά σαφής και η θέση δική μας και αρκετά ασαφής του Συμβουλίου. Γιατί δεν τους πειράζει και τόσο πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε για το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας για να πάρουμε την τελική απόφαση. Θα υπάρξει επιπλέον εφαρμοστική πράξη ή κατεξουσιοδότηση πράξη για τις διαδικασίες, για τις καινοτόμες ενέργειες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι μια συνεχής διαμάχη μεταξύ Επιτροπής και Συμβουλίου. Το Συμβούλιο προτιμάει εφαρμοστικές πράξεις, η Επιτροπή κατεξιοδότηση. Το επόμενο θέμα που θα μας απασχολήσει μεθαύριο είναι το θέμα του τμήματος για την αστική διάσπαση, διάσταση. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για τις επενδυτικές προτεραιότητες και επίσης για το πιο δύσκολο τη θεματική συγκέντρωση που σχετίζεται άμεσα με το γενικό κανονισμό και ενδεχόμενα την πρώτη συζήτηση για τους δείκτες. Οι δείκτες μου είναι εντελώς ακατανόητοι. Η Κομισιόν έχει μια εσωτερική συμφωνία ότι σε κάθε κανονισμό πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ένας κατάλογος δικτών. Αυτή είναι μια οριζόντια αρχή. Οι δείκτες δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τον ε, επιμέρους κανονισμό. Είναι απλώς μεθοδολογία συλλογής στοιχείων. Οι και για τον περιφερειακό και για το Ταμείο Συνοχής κτλ. Είναι ένα τμήμα του νομικού εξοπλισμού του κειμένου. Δεν αρχίσαμε τη συζήτηση για τις τροπολογίες, υπενθυμίζω, γιατί ορισμένοι λένε πως είναι τεχνικό το θέμα. Ορισμένοι λένε ότι πρέπει να το αφαιρέσουμε τον κανονισμό και να το βάλουμε στην ε, εφαρμοστική ή κατεξοδότηση πράξη. Έχουμε τροπολογίες από τους Πρασίνους, από την ΚΟΕ, οι άλλοι δεν υπέβαλαν τροπολογίες. Δεν νομίζω ότι εμείς ως ε, πολιτικοί πρέπει να καθορίσουμε τους δείκτες. Δεν είναι δουλειά μας αυτό. Εμείς πρέπει να καθορίσουμε την πολιτική, όχι τα τεχνικά στοιχεία. Αλλά αν θέλετε να αρχίσουμε τη συζήτηση για τους ε, δείκτες, θα ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας και να δούμε τι θα προκύψει. Γιατί για κάθε κανονισμό θα είναι διαφορετικές οι τροπολογίες. Οι δείκτες πρέπει να δημιουργηθούν από κάτω προς τα πάνω. Ή είναι δείκτες για τη συλλογή στοιχείων που δεν εξηγούν περί τίνος πρόκειται. Αλλά λένε αριθμός ε, χιλιόμετρων, ε, τετραγωνικών μέτρων είναι απόλυτα αναγκαία για τη συλλογή τεχνικών στοιχείων. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι σε ένα νομικό κείμενο. Η Κομισιόν το υπερασπίζεται σαν να είναι θέμα ζωής και θανάτου. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Εμείς έχουμε εντολή να τους απαλείψουμε, αλλά θα δούμε τι θα συμβεί. Ευχαριστώ. Πρώτα η κυρία Ντέλη και μετά θα δούμε. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τι ελπίζω να μπορούσαμε τάχιστα να πετύχουμε τη ε, θέση του Συμβουλίου για πολύ σημαντικά άρθρα σχετικά με τη θεματική συγκέντρωση είτε αυτά τα 5% για την ε, αστική ανάπτυξη γιατί αυτό είναι που αναχαιτίζει τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις. Δεν μας βοηθάει πάντα η Επιτροπή να προχωρήσουμε προς αυτή κατεύθυνση. Τελευταία στιγμή μας δίνει τεχνικά στοιχεία, ενώ για πολλούς μήνες παραμένει σιωπηλή και έτσι αρχίζουμε, ξαναρχίζουμε, ταπώνουμε, βουλώνουμε και θα πρέπει να δούμε λοιπόν και το τίμημα, τι διακυβεύεται, είναι κάτι το πολύ σημαντικό, είναι η ενέργεια. Το θέμα της ενέργειας δεν θα πρέπει να ξεχνάει αυτή την αρμοδιότητα που έχουμε μαζί. Και θα πρέπει να δούμε σε τοπικό επίπεδο τι μπορεί να γίνει. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και κάτι για το οποίο μιλήσαμε σήμερα το πρωί και το γνωρίζω σαν εισηγήτρια και έχει να κάνει με την στέγαση δημόσια και ιδιωτική που είναι τομέας κλειδί για να επενδύσουμε για μια αποτελεσματικότητα ενεργειακή και τις ανώσιμες πηγές ενέργειας. Και στη στέγαση είτε οικοδομή είναι το 40% υπεύθυνο, κατά 40% υπεύθυνο για τα φαινόμενα θερμοκηπίου και θα πρέπει να δούμε την ενεργική αποτελεσματικότητα. Χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ξέρουμε ότι όταν χρησιμοποιούμε επιτόπου το ΦΕΝΤΕΡ, ξέρουμε ότι αποτελεί ένα μοχλό δράσης, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε κάτι παρόμοιο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κορνέλια Κορνέλια παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, ε, Ξεκινώντας, θέλω να πω, πρέπει να προσέξουμε σε αυτούς τους τριμερείς διαλόγους υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές απόψεις, είναι σαφές αυτό. Εμείς πρέπει πολύ προσεκτικά να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της εντολής μας και να μεριμνήσουμε να παραμείνουμε πιστοί στις θέσεις μας και μετά να διαπραγματευτούμε και όχι να επαναχωρήσουμε, να υποχωρήσουμε αμέσω στην πίεση και τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, μια και δεν είμαστε πρόθυμοι να αλλάξουμε την εντολή στα επιμέρους Μέρο σημεία και να μην διαπραγματευτούμε. Ε, πρέπει λοιπόν να μπούμε ακριβώς στο επίκεντρο της υπόθεσης στη μέση και να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, για την πλατφόρμα πόλεων δεν υποστηρίχθηκε καθόλου η πρόταση και στο ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο συμφωνήσαμε δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον βλέπω σε αυτή τη διαδικτύωση αυτά που μας προτάθηκαν δεν είναι η προοπτική να σημειωθεί κάποια πρόοδος. Και στην πρώτη γνωμοδότηση ήδη αναφέρθηκε ότι σε σχέση με αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαμε καταρχήν να έχουμε κάποιο δίκτυο το οποίο θα εντασσόταν, αλλά όχι παράλληλα σε αυτό να χρηματοδοτούνται και άλλες πρωτοβουλίες. Όλα αυτά δεν είναι απόλυτα σαφή και πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση να αποσαφινιστούν. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεύτερο, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και θα δώσουμε προτεραιότητα ή όχι σε μια τέτοια δράση. Έχουμε αρκετά δουλέψει για αυτά και πρέπει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτές τις κατευθύνσεις για την προτίμηση που πρέπει να δώσουμε και να διατηρηθεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό αφορά και την εκπόνηση των προτύπων δράσης. Δεν πρέπει να αφορούν μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και για την τοπική αγορά, τις τοπικές αγορές. Εκεί πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι υπάρχουν συμφέροντα ακόμα και πίσω από αυτό και υλικού χαρακτήρα συμφέροντα. Τώρα προτεραιότητες για τις περιφερειακές ανάγκες που υπάρχουν. Παρόλα αυτά πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε συνέχεια. Είναι ένα σωστό δίπολο που δημιουργείται όχι για την κατάργηση ε, όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής 2020 αλλά κάτι που μπορεί να προσαρμοστεί, να διορθωθεί και να λειτουργήσει και αυτό σωστά. Να συζητήσουμε και την αποδοτικότητα όσον αφορά την χρήση των ενεργειακών πόρων. Σε αυτό συμφωνούμε σε σχέση με αυτά που λένε οι πράσινοι. Δεν έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε πολύ. Πρέπει όλα αυτά να τα κρατήσουμε σε μια δέσμη και να διατηρήσουμε τη θέση μας επ' αυτόν. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανένας να θέλει να παρέμβει. Εσείς θα θέλετε να σχολιάσετε κύριε Όλμπριχτ. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Γενικά νομίζω συμφωνούμε. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι θεμελιώδους χαρακτήρα για μας. Ένα από αυτά είναι η προτεραιότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προτεραιότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λοιπόν Υπάρχει όμως διαφορετική κατάσταση σε σχέση με τα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει αυτό να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικά. Εξακολουθεί να υπάρχει θεματολογικά αυτή η προτεραιότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερο θέμα, η ενεργειακή αποδοτικότητα. Είμαστε ελαστικοί όλοι μας αλλάζοντας, τροποποιώντας τις τιμές όσον αφορά την αποδοτικότητα ενέργειας, αλλά τονίζοντας για τη στέγαση για τα κτίρια, για τις, ε, τα ιδιωτικά διαμερίσματα, την σημασία, τη σπουδαιότητα της ε, ε, αποδοτικότητας χρήσης ενέργειας, ενεργειακών πόρων, διαχωρίζοντας σε σχέση με τα δημόσια κτίρια για παράδειγμα. Το θέμα των διαμερισμάτων των πολιτών είναι έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Μπορεί να δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των ενεργειακών πόρων. Οι πλατφόρμες είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον διότι για τη δική μας κοινοβουλευτική επιτροπή ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται αυτά τα πράγματα από εμά ευθύ εξ αρχής ε, δείχνουν ότι ε, και η Επιτροπή στο τέλος ε, και εκείνη προσαρμόστηκε λέγοντας ότι είναι ένα είδους τεχνολογικό τεχνικού, τεχνικού συντονισμού και συνεργασίας για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας και να δούμε. Θα έπρεπε να είμαστε πιο ανοιχτοί και πιο ελαστικοί συμπεριλαμβάνοντας τη συμμετοχή της, περιφέρειας, της ε, ε, Επιτροπής των Περιφερειών για να διασφαλιστούν αυτοί οι στόχοι ή όχι το επίπεδο της ε, ε, της ε, επέμβαση της Επιτροπής έχει και αυτό τη σημασία του σε σχέση με τα άλλα στοιχεία. Θα έχουμε νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αν πρέπει να αλλάξει η εντολή, ε, φυσικά θα επανέλθουμε στην ε, αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ώστε να αποφασίσει η Επιτροπή σφαιρικά αν συμφωνεί ή όχι με κάποιες τέτοιες αλλαγές. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πολύ σύντομα τώρα να σας ενημερώσω για κάτι όσον αφορά το ETC, τις διαπραγματεύσεις ε, που θα πρέπει να ε, θεωρήσουμε ότι συμπληρωματικά είναι και αυτό πολύ χρήσιμο. Και ένας τριμερής διάλογος ε, συνέβη κατά τα τέλη, χώρα κατά τα τέλη Ιανουαρίου. Γενικά τέσσερις κατηγορίες είναι αυτές που άνοιξαν και εν μέρει έχουμε διαπραγματευτεί επ' αυτών αφορούν και τα θέματα επιλεξιμότητας. Είναι λίγα θέματα πολιτικού καθαρά χαρακτήρα που απομένουν και πρέπει να εξεταστούν κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίασης και μια τεχνικού ε, χαρακτήρα συνεδρίαση που τα αποτελέσματα έχουν ε, υποβληθεί προς έγκριση όσον αφορά την διαπραγματευτική ομάδα. Η κυρία Μάνερ ελπίζει ότι αυτή την εβδομάδα θα είμαστε σε θέση να κλείσουμε τα περισσότερα άρθρα, αν όχι όλα, όσον αφορά τα θέματα υποδιαπραγμάτευση και για τη θεματολογική επικέντρωση και τις προτεραιότητες για τις επενδύσεις υπάρχει στενή διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης και σε σχέση με την ε, τελική συμφωνία δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Ε, αναμένουμε να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ελπίζουμε ότι κατά το Μάρτιο θα καταστεί εφικτό να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο και να προχωρήσουμε στις ε, διαπραγματεύσεις με τις προτεραιότητες. Για θεματική, για τη θεματολογική επικέντρωση υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις ε, όσον αφορά κάποια θέματα εγκρίναμε στην εντολή μας να υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα όσον αφορά προγράμματα ETC προτείνοντας πέντε θεματικές προτεραιότητες αντί τεσσάρων όπως προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει και μια άλλη πρόταση που υποβάλλεται από το Συμβούλιο και που είναι κάπως ε, διαφέρει σε σχέση με την πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου. Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και η Δεσποινής Μάνερ ελπίζει ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια προς εξέβρεση μιας ε, ε, ρύθμισης, μιας λύσης για το μέλλον. Έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, ένα τέτοιο τριμερή διάλογο όπου υπάρχει η πρόθεση να προχωρήσουμε στην εποπτεία, αξιολόγηση, έλεγχο και ε, χρηματοοικονομική ε, διαχείριση θα υπάρξει και η συζήτηση των θεμάτων αυτών στις ε, τεχνικού χαρακτήρα συναντήσεις όπως διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις και σε σχέση με το ETC Αυτά σε σχέση με την ε, ενημέρωση από εσά γι' αυτό την Ευρωπαϊκή ε, Εδαφική Συνεργασία ETC, European Territorial, Territorial Cooperation. Υπάρχει κάποιο που θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ εσεί. Ναι, επαναλαμβάνω την ε, ικανοποίηση όλων όσων συμμετείχαν στον τριμηρή διάλογο για το σε ποιο περιβάλλον διεξάγεται αυτή η συζήτηση. Υπάρχει πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας. Σιγά σιγά όμως προχωράμε κατά την απόψή μας, αλλά τι να κάνουμε και ορισμένα σημεία για την αγροτική ανάπτυξη είναι σημαντικό για μας, για τη συμμετοχή τη χρηματοδοτική όσων θα υποφεληθούν από αυτές τις ενέργειες θα ωφεληθούν και περιμένουμε την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για τον κορισμό του ΦΕΝΤΕΡ και κάτι που συζητήθηκε τώρα τελευταία είναι και η συγκέντρωση γιατί τι προτείναμε στην εντολή πέντε θεματικούς στόχους και το Συμβούλιο το 80% το πήγε σε τέσσερις στόχους και 20% ελεύθερο. Ήταν η πρότασή μας όμως ενδιαφέρουσα, συζητήθηκε αλλά αντίθετα αποφασίστηκε. Λυπάμαι γι' αυτό γιατί είναι διαφορετικές από, από την άλλη περιφέρειες. Χρειάζεται μια κάποια ευληγησία. Και όπως και για τους υπόλοιπους κανονισμούς, πολλά σημεία σημαντικά σε αυτή την ενταφική συνεργασία, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, δεν μας ικανοποιεί πριν από 15 μέρες συμφωνία. Σχετικά με το προπολογισμό ζητήσαμε 7% του προπολογισμού για την εδαφική αυτή ε, συνεργασία και το αναφέραμε σε πολλές εκθέσεις όταν αυτές ε, ψηφιζόνταν ε, στην Επιτροπή μας αλλά μεγάλη απόσταση και όταν είχαμε ακούσαμε αυτά για τα 200 εκατομμύρια νομίζω ότι είμαστε ακόμα μακριά από το στόχο μας αλλά όλοι μας είμαστε πεπισμένοι για αυτήν την εδαφική συνεργασία χρειάζεται να δώσουμε τη μάχη μας στο ο προπολογισμό να είναι ο ανάλογος, ο κατάλληλος ε, και ακόμα για να δούμε αυτή τη διδαυκή συνεργασία ότι μπορούμε να πετύχουμε οικονομία κλίμακος ε, και ανάλογα με το κάθε, την κάθε περιφέρεια δεν είναι σπατάλη χρημάτων. Ε, πολλές σταυροφορίες πρέπει να διεξάγουμε, δύσκολο είναι να πείσουμε και να βάλουμε τα πράγματα πάει στο τραπέζι, πάντα να δίνουμε τη μάχη μας για τον προπολογισμό Πέρα από αυτά, πολλά και διάφορα θα πρέπει να ρυθμιστούν, α πούμε για το ποσοστό σηματοδότηση, πώ τα ποσά υπολογίζονται, διάφορα θέματα που θίξαμε για τα 250 χιλιόμετρα το όριο, για τη συνεργασία τη διαμεθοριακή, το πώ δίδονται αναπρόγραμμα τα χρήματα κλπ. Πολλά και διάφορα που πρέπει ακόμα να συζητηθούν. Τι να σας πω τώρα, που νομίζω ότι εξαντλήσαμε το θέμα. Σας ευχαριστώ. Φρανσουά για το σημείο αυτό για την ευληγησία. Με συγχωρείτε. Τι χειρότερη στιγμή χτυπάει. Πάντα έτσι συμβαίνει. Λοιπόν, ζητήσαμε περισσότερη ευληγησία και τη θεματική συγκέντρωση γύρω από πέντε και όχι τέσσερις στόχους, όπως πρότεινε η Επιτροπή. Το Συμβούλιο της Συμβαστική του Λύσου τι έλεγε τέσσερις ε, θεματικές προτεραιότητες αλλά στο 80% του ποσού και αφήνουμε ε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε λέει ο και 20% για μια ευλίγιστη θέση είναι πως η, η Μαριτερέζ εδώ θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στην Επιτροπή, πώς θα μπορούμε να συμφωνήσουμε, να τα ρυθμίσουμε αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, να ρωτήσω τον Βίκτορ. Μισό λεπτό. Η Τερέσα. Όχι, Ρώσα. Ευχαριστώ. Το Κοινοβούλιο αποδίδουμε σημασία και για τα νησιά τα νησιά που δεν λύθηκε υπόψη ε, αυτά τα 250 χιλιόμετρα για τη διαμεθορική συνεργασία, για τα ποσά που διατίθενται και είδαμε ότι διαγράφεται αυτός αποφάσεις Συμβουλίου. Αυτή είχαμε ζητήσει μέσω της σχετικής έκθεσης Επιτροπής και μέσω του ψηφίσματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2010 και ζητάμε από τόσους διαπραγματεύσεις να προσπαθήσουν ιδιαίτερα για τα νησιά για να, πώς θα αντιμετωπιστούμε στα πλαίσια αυτού του Ταμείου Συνεργασίας. Λαμπέρ. Πολύ σύντομα για την εδαφική συνεργασία. Αν το δει κανείς μακροπρόθεσμα αυτό, τότε το πρόγραμμα αυτό δεν είναι, θα έλεγα, απόλυτα εύληπτο. Διότι βλέπει κανείς ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή κλίμακα όσον αφορά αυτή την εδαφική συνεργασία και τα νησιά συμπεριλαμβάνονται και τα σύνορα τα ξεπερνάμε τις ε, διαχωριστικές γραμμές. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να ε, λειτουργήσει έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε τον νέο στόχο 3, να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει για να ευδοκιμήσει η στοχοθέτηση. Για παράδειγμα, αυτά τα οποία τώρα στο Horizon έχουμε όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, αυτά που καθορίζονται σε αυτό το πλαίσιο. Διαπραγματεύσεις λοιπόν για το Horizon ήταν το πρώτο σημείο και αναφέρθηκε η προσέγγιση της ε, ε, των εξαιρετικών επιδόσεων είναι αυτό που πρέπει να προετοιμάσουμε. Η προετοιμασία για βέλτιστες επιδόσεις ε, μπορούν να γίνουν αυτά μέσω συνεργασίας πανεπιστημιακής συνεργασίας ε, ή συνεργασίας ε, περιφερειών διότι διαφορετικά προς τα πού θα κατευθυνθούμε. Αν όμως από την άλλη πλευρά σκεφτούμε και προβληματιστούμε για τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε, τότε ε, καταλήγουμε στα μέσα και τα εργαλεία τα οποία εδώ και χρόνια αναπτύξαμε για την ε, ε, συνεργασία στο πολιτικό αυτό πλαίσιο. Θα πρέπει να δούμε, χρησιμοποιούμε επαρκώς αυτά τα μέσα για τη διασφάλιση συνέργειας μεταξύ δύο τέτοιων προγραμμάτων. Η περιοχές, οι περιφέρειες της γνώσης, regions of knowledge. Ένα τέτοιο συναφές πρόγραμμα για παράδειγμα, που μεριμνήσαμε τώρα να υλοποιούνται αυτά μέσω των περιφερειακών στόχων που πρέπει να παρακολουθούμε. Αλλά θα πρέπει να δούμε και να ελέγξουμε λειτουργούν όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο του Horizon όπως ε, το θέλαμε με τη νέα πολιτική επενδύσεων που προσεγγίζουμε και υλοποιούμε όλα αυτά λειτουργούν σωστά μπορούν να προχωρήσουν ή τροχοπεδούνται και αποτελματώνονται από τους γραφειοκράτες νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποσαφινιστεί ευχαριστώ ε, yeah, there are some Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις θετικές αλλά και ορισμένες αρνητικές. Πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω ότι ο δεύτερος τριμερής διάλογος θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, 27 Φεβρουαρίου. Και στις 18 Μαρτίου θα διεξαχθεί ο τρίτος και ελπίζω τελευταίος. Αυτό είναι το θετικό. Ευχαριστώ την Κομισιόν και την Ιρλανδική Προεδρία που ήταν διατεθειμένοι να συνομιλήσουν μαζί μας. Αλλά υπάρχουν και λιγότερο θετικές εξελίξεις. Η πιο σημαντική είναι η απόφαση του Συμβουλίου για τις πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές. Γιατί από πλευράς ε, αριθμών ε, ήταν ε, μικρή σημασία στις περικοπές, μόνο δύο δις, το κύριο θύμα της απόφασης ήταν ε, το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Ξέρετε ότι κάναμε μια ιδιαίτερα μακροσκελή κάποιες φορές ανιαρή συζήτηση για το πώς θα πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να γίνει και κατόπιν Σοφρόνος, ιδιαίτερος, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε έναν συμβιβασμό που είπε ότι θα πρέπει να μεταφερθούν δέκα δις από το Ταμείο Συνοχής στο μέσο συνδέοντας την Ευρώπη που θα ανέρχεται λοιπόν σε 40 δις με βάση την πρόταση της Επιτροπής. Αλλά στην τελευταία πρόταση για τις πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές του Συμβουλίου αναφέρονται μόνο 19 δις, λιγότερο από τα μισά δηλαδή. 49% του αρχικού ποσού. Και παράλληλα τα 10 δισεκατομμύρια που επρόκειτο να μεταφερθούν από το Ταμείο Συνοχής Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μας δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα. Γιατί μόνο οι μισές πιστώσεις θα αφαιρεθούν από τα εθνικά συνολικά ποσά του Ταμείου Συνοχής. Αυτή είναι η πρόταση που κάνει το Συμβούλιο. Αυτό δημιουργεί νέα ερωτηματικά. Προφανώς έχει αλλάξει τρομερά η ατμόσφαιρα για το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Διερωτώ με, γιατί κάποια κράτη-μέλη που είχαν δεσμευθεί υπέρ του συνδέοντας την Ευρώπη περιέκοψαν πάνω από το 50% της ε, χρηματοδότησής του. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εμείνουμε στις δεσμεύσεις μας στη συμβαστική μας πρόταση, αλλά θα πρέπει να κάνουμε σκληρές διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για να υποβληθεί μια πιο αξιοπρεπής πρόταση. Επαναλαμβάνω επίσης την πρότασή μας ότι ο κανονισμός ε, του συνδέοντας της Ευρώπης, του κανονισμού, ο κανονισμός συνοχής και ο κανονισμός και όλοι οι κανονισμοί που θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτό το θέμα θα πρέπει να έχουν τις ίδιες διατάξεις. Γιατί αλλιώ δεν πρόκειται να ε, γίνει πραγματικότητα το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη εάν δεν υπάρξουν επαρκείς πιστώσεις. Βεβαίως ε, εδώ ε, αυτό θα δημιουργήσει νέες ανησυχίες και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο άλλα θέματα που θα συζητηθούν. Όπως ακούσατε την προηγούμενη φορά, το Κοινοβούλιο επανυπέβαλε, επανυπέβαλε την πρότασή του για το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Το Συμβούλιο βεβαίως είναι κατά, αλλά ελπίζω στις επόμενες συναντήσεις και το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα δεχθούν να διατηρηθεί το πρόγραμμα αυτό. Επίσης ε, υπήρξε μια πρόταση να εξαιρεθούν ορισμένες ε, δραστηριότητες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Πιστεύω ότι αυτό έχει ε, ξεπεραστεί. Επίσης, για το θέμα της επιλεξιμότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως είπε και ο Γιάνν, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να επιμείνουμε ότι κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να ευνοηθούν για τη χρήση ανανεώσιμων και την ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά όχι οι μόνες. Ε, επιβεβαιώνεται επίσης ε, η χρηματοδότηση αυτών των στόχων για τις κατοικίες. Ανανεώσιμες πηγές δηλαδή και ανανεώσιμες πηγές και ενεργειακή αποδοτικότητα. Το κύριο πρόβλημα για τις δύο επόμενες συναντήσεις θα είναι η συνεχιζόμενη αντίθεση Επιτροπής και Συμβουλίου κατά της ε, ε, υψηλής απόδοσης συμπαραγωγής ε, ενέργειας και θερμότητας και διανομής της. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο τομέας. Σήμερα το πρωί άκουσα όλους τους παρεμβαίνοντες, εισηγητέ, κοιόδης εισηγητέ, την Επιτροπή Περιφερειών και άλλους ε, ενδιαφερόμενους φορείς και ο συναδελφός μου ο Σέρτζο Καρόνα στη γνωμοδότησή του γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η προτεραιότητα και ότι πρέπει να υπάρξουν εδώ προτεραιότητες επενδύσεων. Και ελπίζω να το αποδεχθεί τελικά η Επιτροπή. Πρέπει να ξέρετε ότι το Συμβούλιο μας είπε ότι δεν είναι αναγκαίο αυτό γιατί μπορεί να ανοίξει την πόρτα και για άλλες προτάσεις. Αλλά το Συμβούλιο δεν έκανε καμία σοβαρή συζήτηση για το θέμα αυτό. Ελπίζω την επόμενη φορά να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι, να έχουν σαφέστερη εντολή για να το συζητήσουμε. Αυτά είναι τα κυριότερα προβλήματα για τους κοινού δείκτες. Υποστηρίζω πλήρως τις λογικές προτάσεις του Γιάννου. Ιδιαίτερα διακεκριμένου συναδέλφου και εισηγητού για το Περιφερειακό Ταμείο είναι σαφές ότι αν ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας για να τροποποιήσουμε δηλαδή τους κοινού δείκτες θα δημιουργήσουμε τεράστια προβλήματα ατελείωτες διενέξεις είναι πολύ καλύτερα και πολύ πιο ρεαλιστικά να το επιδιώξουμε αυτό μέσω των εφαρμοστικών πράξεων και όχι να συμπεριλαμβάνεται στο νομοθετικό πακέτο γιατί θα είναι πιο άκαμπτο θα είναι δύσκολο να το προσαρμόσουμε σε ιδιαίτερα μεταβαλλόμενες ε, συνθήκες μέχρι το 2020. Γι' αυτό εμένω στην απλή προσέγγιση που πρότεινε και ο Γιάννη και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι με την πλευρά μας το Συμβούλιο για να κλείσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστούμε εσάς πολύ Βίκτορ. Νίκο, είσαστε ο μόνος σκιώδης εισηγητής παρών. Όχι, δεν θέλετε να παρέμβετε. Κάποιο που θα ήθελε να σχολιάσει ή να παρέμβει για τα μείζωνα θέματα που έθιξε ο Βίκτορ. Λάμπερτ, δεν θέλετε να παρέμβετε. Αν δεν έχουμε κάποιον να σχολιάσει, επ' αυτόν ευχαριστούμε τον Βίκτορα. Ο Ιωακήμ δεν παρίσταται και έτσι δεν πρόκειται να ακούσουμε τα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και από πλευράς του... Α, συγγνώμη, δεν σας είδα εσάς. Παρακαλώ. Νομίζω θα ξεκινήσουμε με το δικό σας σημείο. Είσαστε πρόσδεκτος, παρακαλώ. Ήθελα μόνο να πω δύο λόγια όταν είπατε ότι δεν μπορεί λέει να παραστεί. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τον λόγο. Σύντομα να παρουσιάσω αυτά που στο έγγραφο εργασίας μου για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σκέφτηκα να εκπονήσω και τίθενται υποσυζήτηση. Η αφετηρία είναι οι βιομηχανικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατά το παρελθόν συρρυκνώθηκαν και ουσιαστικά η παραγωγική τους βάση έτυχε μιας φθήνουσας πορείας. Το βλέπουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαλιβουργία, κλωστοϊφαντουργία, παραδοσιακή μηχανουργία ή και εξορρυκτικές δραστηριότητες μεταλλουργικές και άλλες δραστηριότητες σε πολλούς τέτοιους τομείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέμειναν βιομηχανικές έρημοι, βιομηχανικά περιπομένα τοπία και σε σχέση με τα θέματα της έκθεσής μου υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν ως προς όλα αυτά. Σε αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας θέλω να εξετάσουμε τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές και αυτές τις εξειδικευμένες ανάγκες που έχουν αυτές οι περιφέρειες και που είναι και οικονομικού και κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα σε αυτά τα διαφορετικά επίπεδα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι μειονεξίες, τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιφέρειες εξειδικευμένα. Ποιος θα είναι ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Ταμείων, του Περιφερειακού Ταμείου για παράδειγμα μέχρι σήμερα, ώστε για παράδειγμα συγκεκριμένη περιφέρεια που εξετάζω και που θα έπρεπε να δούμε τι μπορεί να γίνει, να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε να παρέμβουμε. Και στον τομέα της περιφερικής πολιτικής και βιομηχανικής πολιτικής, ε, στα όρια τους, η σημασία του βιομηχανικού τομέα θα διαδραματίζει σίγουρα ένα σπουδαίο ρόλο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και ποιες στρατηγικές θα πρέπει να μπορέσουμε να εκπονήσουμε η συνεισφορά όσον αφορά τα διαφθορτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής να δούμε η συνεισφορά τους ποια μπορεί να είναι και η παρουσίαση των προοπτικών σύγκλησης και συνοχής στον τομέα των επενδύσεων. Να έχουμε τα βέλτιστα παραδείγματα για τις διαθροτικές αλλαγές και προσαρμογές. Και τέλος, η σπουδαιότητα αυτής της περιφερειακής πολιτικής από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι αυτών των περιφερειών. Όλα αυτά να τα εντάξουμε σε ένα ολοκληρωμένο, πιο ευρύτερο και σφαιρικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτές τις ανάγκες. Θέματα που συζητήσαμε συζητήσαμε και κατά το παρελθόν και να παρουσιάσω και να δείξω πώς εξειδικευμένα μέτρα όπως η ευφυής εξειδίκευση, smart specialization μπορούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο. Αυτά είναι συντομία ε, για τα θέματα τα οποία εξετάζω στο έγγραφο εργασίας ε, μου και που θα αντανακλώνται και στο κείμενο της έκθεσης. Προσβλέπω στις παρατηρήσεις και σχόλια των συναδέφων. Ευχαριστώ. you very much, uh, Mrs. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εσείς παρακαλώ έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εργασία του και το πρώτο αυτό έγγραφο εργασίας. Επιμένω ότι το θέμα της εκ νέου εκβιομηχάνησης της Ένωσης είναι ιδιαίτερα επίκαιρο γιατί κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι νέα περισσότερα εργοστάσια κλείνουν και αφήνουν στο δρόμο χιλιάδες ε, εργάτες που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθεια εξέβρεσης εργασίας. Η έκθεση λοιπόν αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, μας καλεί να αλλάξουμε λογισμικό να ξεπεράσουμε τους επιδέσμους, να ξεπεράσουμε τις βραχυπρόθεσμες λύσεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ούτω ώστε αύριο η βιομηχανική Ευρώπη να ξαναβρει και πάλι την ευημερία που γνώρισε στο παρελθόν. Ένα πρώτο στάδιο θα πρέπει να είναι ο καθορισμός των τομέων που θα επιδιώξουμε να προωθήσουμε ιδιαίτερα μέσω της ενέργειας των διαφορετικών ταμείων. Πρέπει να δούμε τι έχουν επιτύχει οι ε, βιομηχανίες που προσπάθησαν να περάσουν σε μια οικολογική αναβιομηχάνηση. Υπάρχουν τέτοιοι τομείς όπως ξέρετε που έχουν επιτύχει πολλά, πολλές όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, όλο και περισσότεροι πολίτες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τέτοια προϊόντα που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και που θέλουν να επιδιώξουν να πρασινίσει συνολικά η παραγωγική διαδικασία μέχρι και τη διανομή. Στην εκθεσή σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη την εξάντληση κάποιων πόρων, ιδιαίτερα της ενέργειας. Το κόστος της πρέπει να υποθεί, θα συνεχίσει να αυξάνεται μια βιομηχανική πολιτική πρέπει να λάβει απολύτως υπόψη την ε, εξάντληση κάποιων πόρων. Επίσης, να τονίσουμε ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να παίξουν κύριο ρόλο στη στήριξη αυτής της αναβιομηχάνησης, της οικολογικής αναβιομηχάνησης, πιο οικολογικής και πιο κοντά στους πολίτες. Το πρόβλημα αυτής της αναδιάρθρωσης είναι ότι δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με τη συμμετοχή των εργαζομένων, των μισθωτών. Η νέα βιομηχανική πολιτική πρέπει να υποστηριχθεί από τους μισθωτούς, γιατί αυτοί έχουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και αυτοί θα συνεισφέρουν την ε, προστιθέμενη αξία. Πρέπει να καταδείξουμε ότι πρέπει να συμμετάσχουν, να τη στηρίζουν οι μισθωτοί στα πλαίσια μιας νέας προσέγγισης να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, πράσινες θέσεις εργασίας, τοπικές, που να μην είναι δυνατόν να μετεγκατασταθούν. Πρέπει λοιπόν να καταρτήσουμε τους εργαζόμενους για αυτά τα νέα επαγγέλματα, τις νέες δεξιότητες. Η επαγγελματική κατάρτιση επίσης θα παίξει πολύ θετικό και πολύ βασικό ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί σήμερα να περιοριστεί, να επενδύει απλώς ε, ε, στο συγύρισμα των χώρων μέσω του ΦΕΝΤΕΡ χωρίς να επενδύσει στους ανθρώπους. Πρέπει να επενδύσουμε και στις υποδομές αλλά παράλληλα και στους ανθρώπους. Και όταν λέω ανθρώπους εννοώ όλους τους μελλοντικούς μισθωτούς τα νέα επαγγέλματα και ιδίως τους νέους. Ο ρόλος μας λοιπόν πρέπει να είναι να καταδείξουμε ότι το ΦΕΝΤΕΡ μπορεί ευθύ εξ αρχής να αναπροσαρμόσει τις υποδομές, αλλά συνεργαζόμενοι με το Κοινωνικό Ταμείο που μπορεί να βοηθήσει για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, της ένταξης κτλ, να οθήσουμε τους εργαζόμενους προς τις νέες αυτές ε, κατευθύνσεις, τα νέα επαγγέλματα. Έχει ρόλο να παίξει το Κοινωνικό λοιπόν Ταμείο. Αυτά προτείνω για αυτή την έκθεση λοιπόν. Θα επιθυμούσα η έκθεση αυτή να καταδείξει σε τι βαθμό το κοινωνικό πρότυπο στο οποίο βρισκόμαστε πρέπει να μεταβληθεί γιατί δεν αντέχει άλλο. Η ενεργειακή πόρη δεν είναι ε, άπειρη, είναι πεπερασμένη. Πρέπει να περάσουμε σε ένα νέο τρόπο παραγωγής. Έτσι πρέπει να σχεδιάσουμε την βιομηχανική πολιτική του μέλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέγει η πρόεδρος. Λαμπέρ ώρα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Εδώ ίσως ακούγονται και κάπως διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Πίστευα ότι θα μπορούσα να πω ότι έχω, έχω κάπως απογοητευτεί διότι αντιμετωπίζουμε τη βιομηχανία με μια ας το πω έτσι επικέντρωση στο παρελθόν και σε σχέση με τα βαθιά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες μας θα έπρεπε να είμαστε πιο ισόρροποι στις ε, προτάσεις που υποβάλλουμε. Αν διαβάσετε το έγγραφο για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βιομηχαν... επαναβιομηχανοποίηση που μόλις ε, παρουσιάστηκε, δημοσιοποιήθηκε, μπορώ να πω ότι βλέπω σε σχέση με αυτές τις προτάσεις που παράγονται να λείπουν κάποια πράγματα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ακριβώς όπως αναφέρθηκε και από τη συνάδελφο πιο πριν, ποιο είδους βιομηχανία αναμένουμε και επιθυμούμε και ποια μέσα και εργαλεία χρειαζόμαστε για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Ξεκινήσαμε αυτή ε, σήμερα με τις κρατικές επιδοτήσεις ε, λέγοντας το τι χρειαζόμαστε. Χρειάζονται νέα εργαλεία, νέα μέσα και για τις μεγάλες ε, επιχειρήσεις. Και στη δική μου την ίδια την ε, περιοχή είχαμε μεγάλη, πολύ μεγάλη φθήνουσα πορεία ε, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 και από αυτή την κατάτμιση δημιουργήθηκαν νέες επιχειρήσεις και τώρα έχουμε αυτά τα νέα κύματα για την υψηλού επίπεδου ε, βιομηχάνηση, και βλέπουμε ότι η ε, πολυσχηδής ανάπτυξη ε, διαφορετικών τομέων έχει οδηγήσει σε μια νέα προσέγγιση για το επιχειρήν και την επιχειρηματικότητα για νέους βιομηχανικούς ε, τρόπους δραστηριοποίησης που θα είναι ελκυστικοί. Να δούμε με τη δική μας πολιτική να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις περιοχές εκείνες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα ή να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα και εργαλεία που έχουμε για να ενθαρρύνουμε αυτές τις νέες δραστηριότητες με νέες προοπτικές και στον περιβαλλοντικό τομέα και στο πρασίνισμα της οικολογίας δηλαδή και της οικολογικής δράσης σε όλους τους τομείς της γνώσης και των τεχνολογιών και να δείξουμε και να δούμε πώς μέσα από τους κανόνες και κανονισμούς τέτοιου είδους χρηματοδότηση μπορεί να δώσει μια μελλοντική προοπτική διότι η παλαιότερη βιομηχανική δραστηριότητα που είχαμε στην Ευρώπη δεν βρίσκεται πια εδώ και δεν έχει προοπτικές διότι βρίσκεται το έχει εγκατασταθεί στην Ασία και αλλού. Για παράδειγμα και για την ε, ρομποτοποίηση, αν μπορεί κανείς να ε, μπορέσει χωρίς να πληρώνει μεροκάματα να δημιουργήσει μια τέτοια βιομηχανική δραστηριότητα, ίσως θα υπήρχε μια προοπτική. Να διεξαχθεί μια ευρύτερη συζήτηση λοιπόν επ' αυτών. Και για την ε, ευφυή εξειδίκευση που αναφέρατε, αυτό δείχνει ότι η εξειδίκευση είναι και μια παλαιά αρχή που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να αναπτυχθούν στον οικολογικό τομέα, για παράδειγμα, στον περιβαλλοντικό τομέα. Αυτά θα έχουν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Για παράδειγμα, πολυμορφοποίηση, πολυσχηδείς δράσεις. Φυσικά είναι αναγκαία και η εστίαση, η επικέντρωση για να δημιουργηθεί η ε, κρίσιμη μάζα που θα μπορέσει να οδηγήσει σε ε, θετικά αποτελέσματα. Ίσως λοιπόν προτού υποβληθούν ε, τα συμπεράσματα στην έκθεση, της έκθεσής σας πρέπει να δούμε ποιου είδους βιομηχανία επιθυμούμε και στις συζητήσεις μας θέλουμε να επιτύχουμε. Να ξανασυζητήσουμε λοιπόν για άλλη μια φορά για αυτό το έγγραφο εργασίας προτού καταλήξουμε σε τελικά συμπεράσματα για να μην ακολουθήσουμε μια λανθασμένη κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Uh, anybody else would like to take παίξουμε αν αυτό ήθελε να πει και εκείνη. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψε για ένα έγγραφο εργασίε. άρα μπορούμε να κάνουμε όσε ανταλλαγέ θέλει ο εισηγητή. Αν δεν θέλει κανεί άλλο το λόγο, να ξαναμιλήσει ο κύριο Γκάια Ευχαριστώ πολύ για αυτούς που μίλησαν. Να πω ακόμη ότι η πρόθεσή μου ποια είναι η πρόθεσή μου για αυτή την έκθεση και ποια δεν είναι. Η κυρία Ντέλη λυπάμαι που δεν είναι παρούσα και η συγγήτρια του ΕΛΚ δεν είναι επίσης παρούσα αλλά ο Λάμπερτ Φανίστερλοϊ που την αντικαθιστά είναι παρόν. Να το εξηγήσω λοιπόν. Δεν θα εξηγήσει η έκθεσή μου τι νέε βιομηχανίε θέλουμε. Αυτό θα μπορούσε να το συζητήσει η Ήτρε που είναι αρμόδια για να συζητήσει μια ανακοίνωση της Κομισιόν για βιομηχανική πολιτική που της έχει υποβληθεί. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να συζητήσουμε διαδικασίες και σχέδια, τι θα κάνουμε για τις περιοχές όπως έλεγαν κάποια κείμενα από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες, τι βιομηχανίες να αναπτύξουμε πού κτλ. Και δεν έχω επίσης ε, την πρόθεση να αναφέρω ε, αν οι θέσει εργασία είναι πράσινε, κόκκινε ή μπλε. Στόχο μου είναι να τονίσω ότι έχουμε βιομηχανικές περιοχές στην Ένωσή μας που λόγω της μόνο βιομηχανικής καλλιέργειας που υπήρχε εκεί έχουν συγκεκριμένα μειονεκτήματα. Και υπάρχουν μελέτες που τα καταδεικνύουν αυτά που ασχολούνται με τέσσερις περιοχές της Δυτικής Ευρώπης και από ό,τι ξέρω αυτές οι διαθροτικές αλλαγές ε, αφορούν πρώτα απ' όλα την περιοχή του Ρούρ από όπου προέρχομαι την περιοχή του Μάντσεστα της Λίλ και της Λιέγης είναι λοιπόν ε, βιομηχανικές περιοχές που έχουν κάνει τις αλλαγές που οι χώρες που έχουν μπει πρόσφατα, στην Ένωση ε, δεν τις έχουν κάνει ακόμη. Λόγω λοιπόν της ε, μονομερούς ανάπτυξης υπήρχαν κάποια μειονεκτήματα. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι εκεί ήταν απλώς χειρόνακτες και κάποιοι ήταν ε, manager. Οπότε έχουμε μια οικονομική κατάσταση που δημιουργεί μια δυναμική που δεν επιτρέπει να γίνουν αλλαγές. Παράδειγμα λοιπόν, για ένα συγκεκριμένο μειονέκτημα. Άλλο παράδειγμα, να αναφερθώ και πάλι στην δική μου περιοχή. Δεν είναι δυνατόν ούτε μια τρύπα να ανοίξουμε χωρίς να αντιμετωπίσουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση που έχει να κάνει με δηλητηριώδη υπολείμματα που έχουν αφήσει παλιές βιομηχανίες και επίσης κάποια ερήπια και επίσης και κάποιες ε, βόμβες που δεν έχουν σκάσει από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Πρέπει να καθαρίσουμε αυτές τις περιοχές. Μόνο δημόσιες δαπάνες όμως μπορούν να αξιοποιηθούν. Δύο δυνατότητε λοιπόν υπάρχουν. Είτε θα αφήσουμε αυτές τις περιοχές όπως είναι και θα φυτέψουμε δέντρα ή εάν θέλουμε οποιαδήποτε άλλη ε, βιομηχανική δραστηριότητα θα πρέπει να ε, οικοδομήσουμε τις βιομηχανικές καταστάσεις σε περιοχέ που είναι ακόμη πράσινες και αυτό το θέλουμε. Άρα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες διαδικασίες από πλευράς περιφερειακής και αναπτυξιακής πολιτικής και στόχος μας πρέπει να είναι να διατηρήσουμε την Ένωση. Αν αυτός είναι ο στόχος μας πρέπει να το συνδέσουμε με τα θέματα βιομηχανικής πολιτικής. Αυτό είναι το περιεχόμενο της εκθεσής μου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, θέλετε να πείτε κάτι. Παρακαλώ, να πείτε, να πείτε. Τότε να αλλάξουμε τον τίτλο της έκθεσης, λέει ο κύριος Φανίστελροι να αλλάξει τον τίτλο. Θα μου λύσει το πρόβλημά μου. Πρόεδρος. Κοιτάξτε, το θέμα αυτό Ε, θα μπορούσε ο κύριος Γκάρι να μας κάνει πρόταση και, ο κύριος, ε, και η διάσκεψη των Προέδρων να ε, εγκρίνει την αλλαγή. Περιφερειακές στρατηγικές για βιομηχανικές περιοχές της Ένωσης λέει ο τίτλος. για τις βαριές βιομηχανίες που είναι σε περιοχές που χρειάζονται αναδιάρθρωση. Βεβαίως μπορεί να έχει ενδιαφέρον εκθεσή αλλά θα πρέπει να μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, διμερώς μπορούμε να τα αποσαφηνίσουμε αυτά όταν πρόκειται για παλές βιομηχανικές ε, περιοχές και εστιαζόμαστε σε αυτό. Αυτό ήταν και αντικείμενο της ακρόασης που είχαμε πριν από κάποιες εβδομάδες εδώ και ήταν σχετικά σαφή τα πράγματα τότε. Και αν με αυτά τα οποία παρουσιάζονται, κύριε Φανίστερ Ρόι, δεν ικανοποιώ τις προσδοκίες σας, τότε διμερώς μπορούμε να βρούμε κάποια λύση. Αλλά έχει δίκιο φυσικά η Πρόεδρος επ' αυτού που ανέφερε αν σε σχέση με τον τίτλο που εγώ επέλεξα έχετε άλλες προσδοκίες και δημιουργείται πρόβλημα, ε, τότε ας μην το κάνουμε όλο αυτό. Δηλαδή να ζητηθεί νέος τίτλος με νέα έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Πίσω από αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε δεν είναι η πολιτική αντιπαράθεση πιστεύω. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό που θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε είναι ότι και οι δύο συνάδελφοι μπορούν διμερώς να συζητήσουν τις συζητήσεις τους για να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι προθέσεις και οι στόχοι. Αν υπάρχει ανάγκη για κάποια αλλαγή τίτλου, από ό,τι βλέπω, τότε θα πρέπει το δυνατόν νωρίτερα να μας ενημερώσετε για να αναλάβουμε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες. Γιατί μπορεί να πάρει και δύο μήνες ε, μέχρι να δούμε τι μπορεί να γίνει και ποια θα είναι η έκβαση. Θα είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε το δυνατόν νωρίτερα ειδοποίηση από εσά. Αναμένοντας τώρα την, την εξέλιξη των συζητήσεων την επόμενη φορά όταν θα έχουμε το έγγραφο και θα έχει οριμάσει περισσότερο και από πλευράς έκτασής του, του κειμένου από πλευρά όγκου. Θα τα ξαναδούμε. Σε, την, αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε τώρα τη συνάντηση των συντονιστών. Μετά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι θα έχουμε μια ανοιχτή συνεδρίαση για τους συντονιστές ε, με τα, με, και τα, τους, τα στελέχη του ε, Επιτρόπου Χάν ώστε να μας ενημερώσουν στα αγγλικά για τα αποτελέσματα της ε, Συνόδου Κορυφής. Στις 6.30 θα γινόταν. Αν τελειώσουμε νωρίτερα και θα είναι εδώ γιατί μπορεί να τελειώσουμε νωρίτερα, να είναι εδώ λοιπόν παρόντες για να... Λοιπόν, μέχρι τις 6 και ίσως και νωρίτερα. Okay, so we... Πολύ καλά. Θα ήθελα τώρα λοιπόν οι συντονιστές να παραμείνουν στην αίθουσα για τη συνάντηση των συντονιστών. Και από πλευράς Άλντε δεν υπάρχει συντονιστής από ό,τι μου είπαν. Αν υπάρχει κάποιος πολιτικός σύμβουλος που θα ήθελε να παραμείνει, ευπρόσδεκτος θα είσαστε.